Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην απογευματινή συνεδρίαση. Έχουμε τρία σημαντικά θέματα. Είναι εδώ ο Επίτροπος ε, Σεμέτα για την ε, νέα του πρόταση σχετικά με τον ε, κανονισμό που αφορά στην Όλαφ. Μετά θα συζητήσουμε με τον Βιτόρ Μανουέλ Σίλβα Καλδέρα που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από τη συζήτηση που είχαμε χθε. Και μετά έχουμε την απαλλαγή 2009 που είναι ένα θέμα του κυρίου Χατζημαρκάκη. Μέχρι τις 6 θα συνεδριάσουμε. Από τις 6 και μετά συνεδριάζουν οι συντονιστές. Και για το κάθε θέμα θα αφιερώσουμε μία ώρα. Βλέπω για πρώτη φορά τον δόκτωρα Κέσλερ, τον νέο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ στην αίθουσα. Είναι εδώ, στα, κάθεται εδώ δεξιά. Για πρώτη φορά συμμετέχει στις εργασίες μας. Καλώς ορίσατε κύριε Γενικέ θα συναντιόμαστε σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ελπίζω ότι θα έχουμε ειλικρινείς και ανοιχτές σχέσεις μεταξύ μας για να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ Κοκομπού και της Όλαφ. Πάμε στο σημείο 40 της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Πίτροπε, η Επιτροπή ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα ένα πολύ σημαντικό κείμενο έξω, εκτός από την Ίγκεμπορ Κρέισλερ που είναι έτοιμη με όλες τις τροπολογίες κανένας άλλος δεν κατάφερε μέχρι τώρα να διαβάσει το κείμενο οπότε έχετε το λόγο για την παρουσίαση Thank you very much. ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σύντομα βέβαια το περιεχόμενο της πρότασής μας για τροποποίηση του κανονισμού. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κύριε και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά αυτή που έχω σήμερα. Να σας παρουσιάσω την μεταρρύθμιση του κανονισμού για την Όλαφ στο έγγραφο μελέτης Reflection Paper που σας είχα παρουσιάσει το προηγούμενο καλοκαίρι στηρίχθηκε αυτή η τροποποιημένη πρόταση με ενσωμάτωση των ιδεών και προτάσεων τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. Επίσης, καλύπτονται με την πρόταση αυτή και οι ανάγκες για αναπροσαρμογή του τρόπου εργασίας Ευρωπαϊκής Όλαφ. Η μεταρρύθμιση έχει κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τις αλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της. Ο δεύτερος με τις αλλαγές σχετικές με την υποχρέωση λογοδοσίας από πλευρά της Όλαφ. Ξεκινώ λοιπόν εξηγώντα τι προτείνει η Επιτροπή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανακρίσης της Όλαφ. Κοινό στόχο είναι η βελτίωση τη ε, συνεργασία τη Όλαφ ε, με τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών. Μεταξύ των οποίων βέβαια συγκαταλέγονται και οι δικαστικέ αρχέ. Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει την ανάγκη αυτή τη συνεργασία και τη κρίνουμε σημαντική όχι μόνο κατά την ίδια την ανακριτική διαδικασία, αλλά και για την παρακολούθηση μια υπόθεση ε, μετά τα πορίσματα αυτή τη ανάκριση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, προκειμένου να επιταχύνεται η συνεργασία μεταξύ Όλαφ και αρμοδίων εθνικών αρχών, προτείνουμε να θεσπιστεί μια αρχή, υπηρεσία αύκος ονομάζεται, δηλαδή υπηρεσία συντονισμού κατά της διαφθοράς, που θα προτείνεται από τα κράτη-μέλη, ε, από κάθε κράτος μέλος δεν θα έχει ένα εκπρόσωπο και θα προσφέρει τη συνδρομή της στην Όλαφ, όπως άλλωστε προβλέπεται ήδη και ε, συμβαίνει με τα νέα κράτη-μέλη αυτές οι ε, ανακριτικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υποστήριξη και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όταν διεξάγει ανακρίσεις. Για την παρακολούθηση τώρα των εξελίξεων ύστερα από μια υπόθεση με την οποία έχει ασχοληθεί η Όλαφ, προτείνουμε για την παρακολούθηση να ε, δίνεται η ενημέρωση από την Όλαφ και για να μην επιβαρύνουν υπερβολικά με γραφειοκρατικό φόρτο τα κράτη-μέλη, προτείνεται να ενημερώνουν την Όλαφ κατόπιν δικού της αιτήματο για τη δράση που έχουν λάβει μετά τη διαβίβαση των πληροφοριών της Όλαφ. Για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Οι δε δικαστικές αρχές του κράτου επίση μέλους επίσης θα ενημερώνουν για όποια δράση έχουν το μεταξύ αναλάβει κατόπιν ενημέρωση της, για μια συγκεκριμένη υπόθεση που έχει προσφέρει η Όλαφ. Μια άλλη πτυχή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της έχει να κάνει και με τη βελτίωση της ανταλλαγής ενημέρωσης και πληροφοριών με τα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου όταν υπάρχει προσωπικό μόνιμο ημί ή προϋπολογισμός που έχει αποτελέσει αντικείμενο κάποιας έρευνας, Τη Όλαφ θα πρέπει να δίνουν αμέσω απαντήσει στα ερωτήματα της Όλαφ, ενδεχομένως δεν αναλαμβάνουν και τα προληπτικά διοικητικά εκείνα μέτρα τα οποία θα αποτρέπουν την περαιτέρω ζημία εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προπολογισμού της και θα ενημερώνουν την Όλαφ για ενδεχόμενε νομικές ή πειθαρχικέ ε, διώξει ή μέτρα που έχουν ληφθεί κατόπιν τη υποβολή του πορίσματος τη Όλαφ για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, δυνάμει του κανονισμού, η, Ρόλαβ, η Όλαφ θα έχει ε, προνομή ούχο και ταχύτατη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και την επικοινωνία με τις υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Και επίσης μπορεί να ε, συνάπτει με τη Eurojust, τη Europol ή, τρίτες, ε, ή αρχές τρίτων χωρών διοικητικές συμφωνίες, το ίδιο και με διεθνείς οργανισμούς, Δεδομένων δε των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφιερώνονται στην εξωτερική δράση, θα πρέπει όλα να έχει τη δυνατότητα της συνεργασίας και με τις αρμόδιες αρχές των διεθνών οργανισμών για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της επί τη βάση διοικητικών ρυθμίσεων. Άλλη σημαντικό έργο και πρόκληση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας όλαφ είναι αυτή της ε, επιτάχυνσης των διαδικασιών. Προτείνεται λοιπόν η τακτική επιθεώρηση των διαδικασιών από την Εποπτική Αρχή, η Επιτροπή, και η Όλαφ θα την ενημερώνει σε ποιες περιπτώσεις αποφάσισε να μην λάβει, ε, αναλάβει δράση. Και σε περίπτωση που μια ανακριτική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται μέσα σε 12 μήνων από την εκκίνησή τη, θα πρέπει να ενημερώνει την Εποπτική Αρχή η Όλαφ, την Εποπτική Επιτροπή, για του λόγου ε, ή για τη δράση που έχει αναλάβει κατά εξάμεινα. Ως προς την ε, φύση των εργασιών της, τον τρόπο των εργασιών της, προσπαθούμε να διευκολύνουμε το έργο της με διαφάνεια και ευελιξία, έτσι ώστε να μπορεί ε, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καθηκόντων της. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να δίνει γραπτή εκχώρηση εξουσίας για ορισμένες ε, δράσεις ανακριτικές. Βέβαια παραμένει ο ίδιος επικεφαλής των ανακριτικών ε, δράσεων, δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα όμως είναι και επικεφαλής ενός σώματος το οποίο εγκρίνει το αν θα πρέπει να ξεκινήσει ή να κλείσει μια ανακριτική διαδικασία. Για ορισμένα θέματα, όπως που είχε υπογραμμίσει και το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του, η Επιτροπή προτείνει αυτό να το ενσωματώσει στο εγχειρίδιο των ε, ε, διαδικασιών και όχι στον κανονισμό των ίδιων. Τον ίδιο το ζήτημα της νομιμότητας των ανακρίσεων της Όλαφ. Αυτές οι ανακριτικές διαδικασίες θα πρέπει επίσης να ε, καλύπτονται μέσα από το εγχειρίδιο ε, διαδικασιών που θα εγκριθεί από τον Γενικό ε, Διευθυντή της Όλαφ, ο οποίος θα υιοθετήσει το εγχειρίδιο κατόπιν διαβουλεύσεων με την εποπτική Επιτροπή και τους αρμόδιους φορείς. Προτείνει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία επταετή μη ανανεώσιμη θητεία για το Γενικό Διευθυντή. Δεδομένων δε των πρόσφατων εμπειριών μας προβλέπεται και η θέση του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Σημαντικό θέμα που έχει ήδη συζητηθεί ήταν η αρχή του τεμήνημις για την έναρξη μιας ανακριτικής, μιας ανακρίσεως. Στις εσωτερικές λοιπόν ανακρίσεις ή ε, έρευνες θα μπορεί να αποφασίζει όλα εάν είναι σκόπιμο να παρακολουθήσει μια υπόθεση ε, παραδείγματι παραπομπή της στο IDOC, δηλαδή το ερευνητικό και διοικητικό όργανο της Επιτροπής, ή αντί να την παραπέμψει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Αυτό έχει να κάνει και θα εξαρτηθεί από την φύση και βέβαια τον οικονομικό αντίκτυπο μιας ερευνούμενης πράξης. Η αρχή όμως δεν μήνυμης θα πρέπει όταν εφαρμόζεται να ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες κατευθυντήριε γραμμές που προσδιορίζει και το Συμβούλιο ε, με τα συμπεράσματά του η Εποπτική Επιτροπή δεν θα ενημερώνεται από την Όλαφ για τις περιπτώσεις εσωτερικών υποθέσεων που αποφάσισε να μην παραπέμψει σε κάποια εξωτερική δικαστική αρχή. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στις βελτιώσεις που προσφέρει ως προς την υποχρέωση λογοδοσίας η νέα μας πρόταση. Η πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η εξισορρόπηση, η χρυσή τομή μεταξύ ανεξαρτησίας και λογοδοσίας της Όλαφ. Για να ενισχυθεί λοιπόν η ανεξαρτησία και πέραν της, ε, του διορισμού του Γενικού Διευθυντού για την μη ανανεώσιμη θητεία, η Εποπτική Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθεί να ε, μεριμνά ε, για την πλήρη ανεξαρτησία της Όλαφ κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Και όπως έχει ζητήσει και το Κοινοβούλιο, προτείνουμε να ισχύουν οι κανόνες για την Εποπτική Επιτροπή ε, που, προσ... που, που θα λαμβάνει καθήκοντα από το Δεκέμβριο του 2011. Όσον αφορά το διαρθωτικό διάλογο μεταξύ της Εποπτικής Επιτροπής και των θεσμικών οργάνων για το ανακριτικό έργο της Όλαφ, το Συμβούλιο είχε εκφράσει προτίμηση για μια λιγότερο τυπική προσέγγιση. Το ΔΕ είχε στήσει διαβούλευση μεταξύ των θεσμικών οργάνων με ε, ως αντικείμενο ευρύ φάσμα θεμάτων. Εμεί προσπαθήσαμε πάλι να εξισορροπήσουμε την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό διάλογο για τα θέματα που αφορούν την πάταξη τη απάτη, αλλά και τι ανάγκε για, για ένα τυπικό πλαίσιο με στο οποίο θα εγγραφόταν αυτό. Προτείνουμε ω εκ τούτου ανταλλαγή απόψεων να διεξάγεται τακτικά μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμμετοχή τη Όλαφ και τη Εποπτική Επιτροπή. Η ανταλλαγή αυτή απόψεων θα συμβάλλει στην ε, ανταλλαγή πληροφοριών και βελτίωση συνεργασία των εμπλεκομένων μερών για, ε, με στόχο πάντα τη βελτίωση αποτελεσματικότητα των ε, δράσεων της Όλαφ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει παρέμβαση στις ανακριτικές της, ε, στις υποθέσεις της, στις έρευνές της. Μέχρι στιγμής λοιπόν ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διαδικαστικές εγγύσεις για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις ανακρίσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε με μεγάλη προσοχή το ζήτημα της προστασίας αυτών των δικαιωμάτων, ε, των διαδικαστικών δικαιωμάτων, των δικονομικών δηλαδή δικαιωμάτων. Πρέπει να καταστούν όμως πολύ πιο σαφή και διαφανή και να ισχύουν για κάθε έρευνα της όλα τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική ανακριτική δράση. Αυτές οι δικονομικές εγγυήσεις ε, σημαίνουν σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως θα αναγνωρίζει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές λοιπόν ανακρίσεις, τα δικονομικά δικαιώματα καλύπτονται από την τροποποιημένη μας πρόταση. Το δικαίωμα του ε, υποκειμένου της ανακρίσεως σημαίνει ότι δεν αναφέρεται το όνομά του Σημαίνει επίση ότι ενημερώνεται συνοπτικά για τα πραγματικά γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο τη ανάκριση, ότι έχει το δικαίωμα να κάνει σχόλια, ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή κάποιου ανθρώπου, ε, προσώπου τη επιλογή του κατά την ε, ανακριτική διαδικασία ή την λεγόμενη συνέντευξη, ότι έχει δικαίωμα χρήσης μιας από τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά επιλογή και επίσης ε, την αρχή ότι κάθε υποκείμενο ανακρίσεως έχει το δικαίωμα να αποφύγει ε, κάποια δήλωση η οποία θα τον ενέπλεκε, θα τον την ενέπλεκε περισσότερο θα τον ενοχοποιούσε. Όλα αυτά πιστεύουμε θα πρέπει να καταγραφούν στο εγχειρίδιο των διαδικασιών της Όλαφ, όπως θα εγκριθεί αυτό από το Γενικό Διευθυντή. Και επίσης θα πρέπει να εγγραφούν στο πλαίσιο των ανακριτικών διαδικασιών που αναπτύσσει ο Όλαφ ακόμη και σε αυτές που έχουν διοικητικό περισσότερο χαρακτήρα. Η ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί και στο δικαίωμα της ε, προσφυγής, ε, δηλαδή μέλος του προσωπικού ή ε, του διεθνού προσωπικού που αποτελεί υποκείμενο μιας ανάκρισης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μια ανεξάρτητη γνώμη σε σχέση με την, με την προστασία των δικονομικών του δικαιωμάτων. Αυτό πάντα με την επιφύλαξη της, ε, του δικαστικού ελέγχου από το πρωτοδικείο του Λουξεμβούργου. Η διαδικασία της προσφυγής πρέπει να προβλεφθεί από τον Γενικό Διευθυντή και το επιτελείο του και να εγγραφεί στο εγχειρίδιο των διαδικασιών, το εγχειρίδιο λειτουργίας όλων. Ταυτόχρονα με την λειτουργία της Εποπτικής Επιτροπής και προκειμένου να ε, αποφευθούν επικαλύψεις έργου θα γίνεται η εξέταση της προσφυγής αυτής κατά τρόπον απόλυτα ανεξάρτητο. Το δε επιτελείο του Γενικού Διευθυντή θα δίνει απαντήσεις ως προς τα μέτρα ε, που ελήφθησαν για την ε, θέση λειτουργίας της διαδικασίας προσφυγής και τα εξέτασέ Κυρίε και κύριοι, ε, προσπάθησα εν συντομία να δώσω απαντήσεις στα θέματα που καλύπτει αυτή η αναθεώρηση του κανονισμού μας. Ελπίζω ότι είναι ικανοποιητική η έκθεση και πάνω απ' όλα ότι ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα του Κοινοβουλίου όπω τα είχατε εσεί καταθέσει στο παρελθόν. Πιστεύω ότι έχουμε ε, υποβάλει ρεαλιστικές και πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Σόλαφ. Εδώ βλέπετε πιστεύω να αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό ε, το σύνολο των ετοιμάτων για βελτίωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στηρίζομαι στη δική σας ε, συμβολή για έναν επικοδομητικό διάλογο και βελτίωση περαιτέρω της προτάσεως με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων μέχρι το τέλος του 2011. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Επίτροπε Σεμέτα. Η συνάδελφος Γκρέσλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θέλω να χαιρετήσω και τον νέο διευθυντή της Όλαφ για να τον συγχαρώ για τη νέα θέση του. Στο δύσκολο έργο του του, έχω, του εύχομαι κάθε επιτυχία. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω για το έγγραφο εργασία. Χρειάστηκε 1,5 χρόνο για να μπορέσουμε να το έχουμε στα χέρια μας. Και αυτό το έγγραφο εργασία το οποίο ζητήσαμε και το οποίο έχει, κάνει κάποιες, ε, έχει τροποποιηθεί σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο είναι πράγματι μια τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν. Χαίρομαι λοιπόν για τον διάλογο που είχαμε και για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία συναπόφασης που μας εμπλέκει με το Συμβούλιο. Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρεξήγηση σε σχέση με το θέμα της συναπόφασης. πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία σε μια περάτωση. Έχουν περάσει δυόμιση χρόνια σχεδόν. Εγώ δεν νομίζω λοιπόν ότι έχουν προχωρήσει αρκετά γρήγορα τα πράγματα. Πάντω, είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ένα έγγραφο εργασία, το να υπάρχει ένα έγγραφο εργασία μεταφρασμένο σε όλε τι γλώσσε, το οποίο να εκτιμά το κείμενο τη Κομισιόν και να περιλαμβάνει τι τροπολογίε μας επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία τον Νοέμβριο του 2008, θέλω να σα υπενθυμίσω ότι ήταν αυτά που είχαμε ζητήσει τότε το Νοέμβριο του 2008. Ο στόχο αυτή τη μεταρρύθμισης μέσα στα πλαίσια τη Κομισιόν ήταν να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία, καλύτερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τη Όλαφ και των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Eurojust, τη Europol και όλων των άλλων ε, φορέων και των μελλοντικών τότε φορέων που θα προέκυπταν από τη Σύνθηκη τη Λισαβόνα και ο στόχος ήταν η Κομισιόν να διευκολύνει και τις σχέσεις μεταξύ Όλαφ και κρατών μελών, ώστε οι έρευνες της Όλαφ στα κράτη-μέλη να μπορέσουν να καταλήξουν σε καλύτερα αποτελέσματα χάρη σε μια καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Οι στόχοι λοιπόν της Όλαφ και του Γενικού Διευθυντή της θα έπρεπε να γίνουν σαφέστεροι και θα έπρεπε να υπάρχουν και απαραίτητοι πόροι οποίοι στην που θα το εξασφάλιζαν αυτό. Επίση υπήρχε και η ανάγκη να υπάρχει καλύτερο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων στο βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Το ερώτημα είναι κατά πόσο λοιπόν επετέθησαν αυτοί οι στόχοι. Το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα ήθελε να υπάρξει μια διαβούλευση, όπως αυτή που γίνεται σε επίπεδο νομοθετημάτων, ώστε σε περιπτώσεις που λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της απάτης να υπάρχει μια κοινή δράση των δύο θεσμικών οργάνων αυτών. Επίσης, προτού λυθούν μέτρα από την πλευρά της Όλαφ, διοικητικού χαρακτήρα μέσα δηλαδή, θέλαμε να υπάρχει άμεσα πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Όλαφ προς τα θεσμικά όργανα σε σχέση με την πορεία των ερευνών και ο στόχος μας φυσικά ήταν σε τελική ανάλυση να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις απώλειες κονδυλίου. Επίσης θέλαμε να έχουμε καλύτερη σύνδεση με την Eurojust και την Europol και να έχουμε ευκολότερη ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης να καταλήξουμε και συμφωνίες με τρίτα κράτη για συνεργασίες σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απάτης ή γενικά σε περιπτώσεις που θα πρέπει να διεξαχθούν ανακρίσεις. με ανάμεικτο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, έλαβε υπόψη την, τις προτάσεις αυτές ε, η Κομισιόν ε, και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι εμείς καταθέσαμε 220 τροπολογίες από τις οποίες πέρασε ένα σχεδόν 60% στην Ολομέλεια. Το πρώτο πακέτο θεμάτων που μας απασχόλησε ήταν το θέμα της συνεργασίας με τα άλλα θεσμικά όργανα ξεκινώντας από την ανταλλαγή πληροφοριών. Μεταξύ των οποίων μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει παραμένει σε ένα πολύ γενικό επίπεδο. Πιστεύω ότι η Κομισιόν εδώ έχει περιορίσει και τη συμφωνία της με τη Eurojust και τη Europol και παραμένει σε ένα επίπεδο υποδέστερο από αυτό που είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με γενική συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων να κάνει η Κομισιόν για την συνεργασία με αυτού του φορεί. Και έτσι θα πρέπει να επανέλθουμε πιστεύω σε όλα αυτά τα θέματα γιατί ιδίω μέσα στο νέο πλαίσιο το οποίο δημιουργεί η συνδίκη τη Λισαβόνα θα πρέπει να διαλευκαθεί καλύτερα ή θα πρέπει ακόμα και να αναδιατυπωθεί ο ρόλο τη Όλαφ. Ένα δεύτερο σημείο αφορά τη σχέση της Όλαφ με τα κράτη-μέλη. Εδώ η θέση του Κοινοβουλίου ήταν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίδουν ένα, μια έκθεση ε, follow-up, μια έκθεση συνέχεια σε σχέση με τις διαδικασίες τις ερευνητικές και ανακριτικές που λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη. Σας πενθυμίζω ότι οι στατιστικές που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι μόνο 7% των διαδικασιών καταλήγουν κάπου και τα άλλα 93% καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο να ξέρει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγο καλύτερα ποια είναι η διαδικασία η οποία γίνεται στα κράτη-μέλη. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν και εθνικά σημεία επαφής για τις διαδικασίες της Όλαφ και θέλαμε επίσης οι διαδικασίες αυτές να οδηγούν σε διαβούλευση σε τακτικό επίπεδο με το, με το Συμβούλιο. Η Κομισιόν δέχτηκε την ε, θέση μας να υπάρχουν εθνικά σημεία επαφής, αλλά για την έκθεση που πρέπει να μας δίνουν τα κρατημέλη σε σχέση με τις έρευνες, αυτό το απέρριψε και απέρριψε και την ιδέα της ε, διαβούλευσης με το Συμβούλιο. Αν θέλουμε όμως εμείς η ΟΛΑΦ να λειτουργήσει σε μια αποδοτική βάση, πιο αποτελεσματική βάση στα κράτη-μέλη, τότε αυτό είναι μια απαράγραπτη ανάγκη να έχουμε τα σημεία επαφής και την, ε, τις σχέσεις τις εκθέσεις ε, για τη συνέχεια. Ένα περαιτέρω στοιχείο αφορά το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ε, ΟΛΑΦ. Η κάλυψη αυτής της θέσης με μια προκήρυξη διαγωνισμού με ειδικά προσόντα για τους υποψηφίους και φυσικά που να περιλαμβάνουν μια καλή γνώση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό ήταν μια διεκδίκηση του Κοινοβουλίου είχαμε ζητήσει να γίνεται δημοσίευση για εννέα μήνες τουλάχιστον και να υπάρχουν τρεις μήνες για την επιλογή των ε, τελικών υποψηφίων και προβλέπαμε να γίνει πέντε χρόνια η θητεία του Γενικού Διευθυντή με, περίοδο, με δυνατότητα μίας ανανέωσης και μόνο. Και είχαμε επίσης ε, προβλέψει να υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς και ένας κώδικας διαδικασίας μέσα στην Όλαφ και να υπάρχει η δυνατότητα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος και σε αυτές τις περιπτώσεις. Για την διαδικασία αυτή η Κομισιόν δεν έδωσε συγκεκριμένες ε, λεπτομέρειες και θέσεις. Είπε ότι αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί στη διαβούλευση. Ε, προέβλεψε μια διαδικασία εξάμηνη για, την, ε, για τον διαγωνισμό, για την προκήρυξη του διαγωνισμού, για τη διάρκεια του διαγωνισμού. Έλαβε υπόψη επίσης την ανάγκη το προφίλ του ε, υποψηφίου να έχει αυτό το χαρακτήρα που ζητήσαμε, αλλά η διάρκεια της θητείας είναι 7 έτη κατά την Κομισιόν. Και θα πρέπει ο Διευθυντής να δίδει μια έκθεση πεπραγμένων ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. και κάτι το οποίο επίση χαιρετίζω, προβλέπεται να υπάρχει ένα ένας αναπληρωτής γενικός διευθυντής. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητε του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να συμβουλεύεται ένα εσωτερικό σώμα, ένα διοικητικού συμβουλίου προτού προχωρήσει σε δίωξη, σε άνοιγμα διαδικασίας. Υπάρχει τώρα ένα είδος εγχειριδίου, εγκολπίου, αλλά αυτός δεν είναι ο κώδικας συμπεριφοράς ο οποίος θα μας προσέδιδε μια μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και γι' αυτό πιστεύω πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και η δυνατότητα αυτο, αυτεπάγγελτης παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει ληφθεί υπόψη στην πρόταση της Κομισιόν. Μπορούμε να είμαστε λοιπόν εν μέρη ικανοποιημένοι για ορισμένα σημεία, αλλά για άλλα σημεία θα χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση με την Κομισιόν αλλά αυτό το οποίο για μας είναι το πιο σημαντικό είναι η σημαντική συμμετοχή του Κοινοβουλίου για την επιλογή των υποψηφίων. Αυτό είναι κάτι στο οποίο εμεί πιστεύω θα πρέπει να επιμείνουμε. Το πέμπτο σημείο είναι τα δικαιώματα των εμπλεκομένων στις διαδικασίες αυτές και οι διαδικασίες. Η έννοια του review advisor, δηλαδή κάποιο ο οποίος θα μπορούσε να κάνει μια εποπτεία της διαδικασίας αυτής και αυτό έχει εξαφανιστεί από το κείμενο της Κομισιόν που ήταν ένα αίτημα του Κοινοβουλίου και στη θέση του το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να δίνει εντολή σε ένα άτομο να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στα πλαίσια της Όλαφ αλλά δεν, είναι, δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώ ο ρόλο αυτού του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια τη Όλαφ και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επανέλθουμε. Αυτά τα οποία επίση συζητήσαμε να υπάρχουν υπομορφή δικονομικών εγγυήσεων για την ε, για την ε, ενότητα της ε, ανακριτικής διαδικασίας αυτό δεν ε, έχει εξασφαλιστεί. Δηλαδή οι εθνικοί ανακριτές δεν υποχρεωμένοι να δεσμεύονται με την ίδια διαδικασία που θα ακολουθεί η Όλαφ. Και αυτό το σημείο επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί από την Κομισιόν. Εμείς είχαμε αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική διαδικασία ώστε να μπορούμε καταρχήν να ξεκαθαρίζουμε τα θέματα αυτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία μέσα στην ΟΛΑΦ, αυτό έχει εξαφανιστεί επίσης από την πρόταση της Κομισιόν. Επίσης και η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει, έχει εξαφανιστεί. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος της νομιμότητος επίσης είναι κάτι το οποίο χρειάζομαι, χρειάζεται να υπάρχει σε μια συγκεκριμένη μορφή. Θα πρέπει όμως να υπάρξει και μια διαδικασία εδώ για να προστατεύεται η Όλαφ από δυνατές παραβιάσει της νομιμότητας. Εν κατακλείδη λοιπόν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε επιτύχει, όπως παραδείγματος χάρη τα θέματα αυτά της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια συζήτηση με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Εγώ έχω καταθέσει το έγγραφο εργασία, όπου περιλαμβάνω τα στοιχεία τα οποία δέχτηκε η Κομισιόν και τα οποία δεν δέχτηκε και επί τη βάση αυτή μπορούμε να κάνουμε μια περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ συνάδελφος Μπάλτσιτης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αρκετά δύσκολο να παίρνει κανείς το λόγο μετά την κυρία Γκρέσλε, διότι είπε ό,τι έπρεπε να πει κανείς. Σημειώσαμε κάποιες ε, παρατηρήσεις, εγώ είχα σημειώσει κάποιες παρατηρήσεις που έλεγα να προτείνω στην ε, Κομισιόν, αλλά καλύφθηκα. Όπως σωστά υπόθηκε, όταν συζητάμε για τον ρόλο της Επιτροπής Εποπτείας και το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι υπόλογος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να γράφονται καθαρά και ξαστέρα στα έγγραφα. Η δυνατότητα προσφυγής κατά των ε, δραστηριοτήτων ε, της Όλαφ, η ανταλλαγή πληροφόρησης, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στα κράτη μας έχουμε διαφορετικά συστήματα μεταξύ τους ακόμη και μέσα σε μια ίδια χώρα όλα αυτά τα θεσμικά όργανα δεν καταφέρνουν να μιλούν μεταξύ τους και πρέπει να, τα να οργανώνονται όλα αυτά σε ένα ανώτερο επίπεδο. Τα πρακτικά. Ο απολογισμός επίσης είναι κάτι το σημαντικό, το να δίνει κανείς λόγο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Πρέπει να διασφαλίζουμε εμείς όλους τους απαραίτητους όρους στην Όλαφ να εργάζεται αποτελεσματικότερα να προχωρά με μικρά βήματα και ελπίζομαι ότι στην αρχή των εργασιών μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ευωδώσει η αλλαγή, η αλλαγή, να ευωδώσουν οι αλλαγές στα πλαίσια της Όλαφ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις πληροφορίες του. Και εγώ τώρα θα επανέλθω στις εγγύησει και στα δικαιώματα των ελεγχομένων από την Όλαφ Δηλαδή, εντάξει, ο κάθε γενικός διευθυντής ε, καλό θα ήταν να βγάζει το εγχειρίδιό του, αλλά δεν μιλάμε για την φύση αυτού του εγχειριδίου που θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν, δεοντολογικό, έναν κώδικα δεοντολογίας ε, έναντι των ελεγχομένων. Και αυτές ε, οι εγγύσει είναι πολύ σημαντικές. Εδώ δίνεται ένας κατάλογος για το τι πρέπει να κάνει κανείς μέσα στο εγχειρίδιο σύμφωνοι, αλλά δεν υπάρχει ένας κώδικας, ένας κώδικας που να διασφαλίζει ιδεοντολογικά και τους ελεγκτές και τους ελεγχόμενους. Θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο πώς ε, θα καλύψουμε αυτήν την αδυναμία. Και αυτό που έλεγε και η συνάδελφος η κυρία Γκρέσλε για τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή. Το είδαμε κατά τον διορισμό σας. Θέλω να ρωτήσω στον Επίτροπο. Τι ρόλο προσδίδει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς στο παρελθόν είχαμε μια αρκετά αρνητική και φλού κατάσταση που αποδυνάμωνε που αποδυνάμωνε τον διορισμένο διευθυντή διότι έβρισκε ένα όργανο έβρισκε ανοιχτή μια πολεμική με ένα όργανο Λοιπόν, πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται από την σύγκρουση μεταξύ θεσμικών οργάνων. Η κυρία Αντριάσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μια σύγκριση μεταξύ Δεκεμβρίου του 10 και Μαρτίου του 2011 του οργανογράμματος δείχνει ότι έφυγαν τρεις από την ε, ε μονάδα για τα κατά ταμεία. Γιατί? Γιατί έχασε τρεις υπαλλήλους αυτή η μονάδα που έχει το υψηλότερο, σημαντικότερα προβλήματα στους τελευταίους λογισμου. Το 2006 η Επιτροπή δημοσιεύει τελευταία της πρόταση για την μεταρρύθμιση της Όλαφ. Το Κοινοβούλιο υιοθετεί με 100 περίπου τροπολογίες το ψήφισμά του Μπορεί η Επιτροπή να μας δείξει σαν να πίνακα ποιες τροπολογίες έλαβε υπόψη, ποιες απέρριψε και για ποιους λόγους. Το νέο άρθρο 9,7 δίνει του κανονισμού δίνει στην όλα αρκετές, αρκετές ε, δυνατότητες για να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί την τελική της έκθεση σχέση με τον ε, ότι είναι αναγκαίες, αναγκαίοι όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Κύριε Στάση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ από τη δική μου πλευρά να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και για τις εξηγήσει που έδωσε. Για τα αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε τώρα. Το 2007-2008 το Κοινοβουλίο μας επενέδισε πάρα πολύ ενέργεια στις πρώτες αυτές προτάσεις είχαμε καταφέρει να ξεπεράσουμε τις στενές παραταξιακές γραμμές και να συνεργαστούμε μεταξύ μας και δώσαμε στην Επιτροπή, στον τότε Επίτροπο, πάρα πολύ σημαντικές τροπολογίες για τα θέματα αυτά. Εγώ έχω εδώ πέρα στο διαδίκτυο την, τη συζήτηση της 20 Δεκεμβρίου ξαναάκουσα τα στοιχεία αυτή της συζήτησης και μετά από αυτά που είπε και η κυρία Γκρέσλερ, βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλες αποστάσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε τότε ζητήσει. Πρέπει λοιπόν να καταθέσουμε ακόμα τροπολογίες για να εξασφαλίσουμε την, ε, μεταξύ άλλων την εμπιστευτικότητα των δημοσιογραφικών πηγών να εξασφαλίσουμε επίσης μια καλύτερη προστασία αυτών οι οποίοι καταγγέλουν κάποια ατασταλία ή απάτη. Και αυτό ήταν μια τροπολογία που είχε υποστηρίξει το Κοινοβούλιο μας. Ανοιχτό πνεύμα και διαφάνεια στις πληροφορίες που δίνονται στο ευρύ κοινό, στην κοινή γνώμη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν αντανακλώνται στην τωρινή θέση της Κομισιόν. Βέβαια θα πρέπει να τα ξαναζυγίσουμε όλα αυτά γιατί δεν έχουμε διαβάσει πλήρως το κείμενο αλλά έχει δίκιο η κυρία Αντρέσεν όταν ζητάει να υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο σύνοψη των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της τύχης την οποία, ε, της οποίας έτυχαν μετά. Εγώ θα ήθελα να ξέρω γιατί ορισμένε τροπολογίε ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απερίφθησαν. Δεν λέω ότι δεν έχει το δικαίωμα το κάνει η Κομισιόν, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αιτιολόγηση. Γνωρίζοντας την κυρία Γκρέσλε, ξέροντας ότι είναι μια διαδικασία συναπόφασης, ξέρω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο και νομίζω θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρουσιάσατε ένα νέο σχέδιο κανονισμού για την Όλαφ. Ο κύριος Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση. Εγώ θα υποστήριξω τόσο από κύριο Στάς όσον αφορά την απογραφή των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Δηλαδή της εφαρμογής τους. Θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό ελήφθη υπόψη ε, η άποψη του Κοινοβουλίου στην τροποποίηση αυτή. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με την ανεξαρτησία και με την απαγόρευση ανανέωση της θητείας ε, και με τη διάρκεια βέβαια της θητείας που είναι αντιθέτες με τη δική μας πρόταση. Εμείς είχαμε ζητήσει από ε, δύο θητείες πενταετής. Εσείς ορίζετε μία επταετή, μία ανανεώσιμη. Γιατί. Δεύτερον. Η σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας θα πρέπει να κάνουμε δεκτές τις διαφορές αν Δεν μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχουν αυτές τις διαφορές. Ευχαριστώ, Γκρέσλε. Ναι, Πρόεδρε, με συγχωρείτε που ζητώ και πάλι το λόγο. Έχω τρει σημαντικέ παρατηρήσει. Καταρχά, το θέμα των δημοσιογραφικών αυτών πηγών των πληροφοριοδοτών που ακούστηκαν νωρίτερα. Δεύτερον, την τροπολογία περιθμών 40 ω προ την πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα τη Όλαφ. Ε, που όμω δεν έγινε δεκτή, δεν σωματώθηκε στο κείμενο. Και φαίνεται ότι αυτή η πρόσβαση για άλλη μια φορά, την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα, ε, αποκλείστηκε. Βλέπουμε λοιπόν ότι για το Γενικό Διευθυντή προβλέπεται στο νέο έγγραφο να καταθέτει γραπτός ε, υποδείξεις προς, τους, προς το προσωπικό του. Εάν λοιπόν ε, δίνει τέτοιου είδου υποδείξει. Εμεί δεν θέλουμε να, να πλήξουμε το κύρο αυτού του θεσμού. Αλλά όταν ο ίδιο ο Γενικό Διευθυντή δώσει ε, εντολέ γραπτέ και αυτό ορίζεται και στην νομοθεσία και στη συνέχεια είναι παράνομε οι εντολέ που δίνει και παρεμβαίνει το δικαστήριο. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί να υποπέσουμε σε τέτοιο σφάλμα. Στα 4849, πάλι ε, στο ζήτημα τη εξίσωση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών και στα δικαιώματα του ε, υποκειμένου της ανάκρισης. Είναι καλύτεροι δηλαδή οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύτεροι άνθρωποι, είναι αναμφίβολο ότι ε, διαπράττουν λιγότερα δικήματα, θα έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική συνένεση ότι ο στόχος μας είναι να δεχτούμε φυσικά το ότι μπορούν να υπάρχουν εσφάλματα, αλλά να φτάσουμε σε ένα μηδενικό επίπεδο απάτη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για αυτά τα οποία μας παρουσίασε. Τώρα, σε επίπεδο ενιολογικό, η έννοια του οργανισμού, του οργάνου και του θεσμού. Επειδή αυτές οι έννοιες επανέρχονται πάρα πολλές φορές, καλό ήταν στο σημείο 2 που υπάρχουν ορισμοί να έχουμε καλύτερους ορισμούς. Το ελεγκτικό συνέδριο παραγωγής χάρη. Πώς εμπίπτει μέσα στους ορισμούς αυτούς. Επίσης, τις ανταλλαγές πληροφοριών. Είναι πάρα πολύ ασαφείς οι έννοιες που χρησιμοποιούνται. Λέμε μια διοίκηση μπορεί να πληροφορήσει την ΟΛΑΦ, η ΟΛΑΦ μπορεί να δώσει σε κάποια διοικητική αρχή κτλ. Όλα αυτά όμως δεν είναι αρκετά επακρίβη. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την ε, απάτη, δεν γίνεται αυτό μόνο με καταγγελίες, γίνεται και με ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένους όρους, απόλυτα συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι θα υποχρεώνουν όλους αυτούς που έχουν πρόσβαση στην ε, δημόσια σφαίρα και στην διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και εδώ σκέφτομαι συγκεκριμένα το ελεκτικό συνέδριο αλλά και τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια τα οποία στα πλαίσια των ελέγχων τους μπορεί να αποκομίσουν πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση της απάτης. Οι ορκωτοί λογιστές, παραδείγματο χάρη, επίση οι οδηγητικοί φορείς, λογιστικοί φορείς που μπορούν να κάνουν κάποιες, ε, κάποιους ελέγχους στους ε, αποδέκτες ταμείων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να βρουν πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες. Θα είναι λοιπόν χρήσιμο να καθορίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να δώσουν πληροφορίε προ την ΟΛΑΦ, η οποία ΟΛΑΦ μετά τι αξιολογεί και κάνει τη δουλειά τη. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπο Εμέτα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ <clears throat> για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας. Είναι γεγονός ότι υπήρξε αρκετά μακροχρόνια η διαδικασία. Εγώ όμως, όπως ξέρετε, ξεκίνησα τις, ε, ε ανέλαβα τις ευθύνες μου μόνο το Φεβρουάριο του 2010. Και από τη στιγμή αυτή έκανα ό,τι μπορούσα, σας έδωσα το έγγραφο προβληματισμού που ζητήθηκε από την Επιτροπή σας και σήμερα έρχομαι με την τροποποιημένη πρόταση για τον κανονισμό για την ΟΛΑΦ όπως ε, ζητήθηκε και από την Επιτροπή σας. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρήσουμε ένα καλό πνεύμα συνεργασίας γιατί πιστεύω ότι και ο στόχος μας είναι ένας κοινό στόχος να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της Όλαφ και να άρουμε τα προσκόμματα τα οποία ενδεχομένω υπάρχουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ε, Όλαφ. Οι οι βουλευτές της Επιτροπής έχουν θίξει πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν θα μπορέσω μάλλον να τα αντιμετωπίσω όλα πλήρως. Θα πρέπει να επανέλθουμε στη συζήτηση και αργότερα. Συμφωνώ με την ε, κυρία Γκρέσλε ότι η διαδικασία αυτή συναπόφασης είναι μια καλή αντιμετώπιση και εμείς φυσικά από τη δική μας πλευρά την έχουμε σεβαστεί απόλυτα. Αλλά στα πλαίσια της προετοιμασίας της οριστικής απόφασης θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, να κρατήσουμε ένα θετικό διάλογο και να <clears throat> συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Για τα κύρια τώρα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν, για τις ε, <clears throat> διαθεσμικού χαρακτήρα συμφωνίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε μια σαφέστερη μνήα αυτών των συμφωνιών που έχουν γίνει με τη Europol και τη Eurojust. Και όπως ξέρετε η Όλαφ έχει ήδη μια συμφωνία με τη Eurojust για πλήρη συνεργασία και δεν βλέπω να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην συγκεκριμένη αυτή μορφή συνεργασίας. Για τα θέματα αυτά τα οποία επίσης αναφέρθηκαν για ένα διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των θεσμικών αρχών, μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και η δική μου κατανόηση είναι ότι αυτό το οποίο έχουμε προτείνει ως Κομισιόν είναι μια καλή συμβαστική λύση η οποία θα επιτρέψει την διατήρηση της λογοδοσίας της Όλαφ προς, το, προς τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, αλλά συγχρόνως διατηρώντας και τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε πιο ευέλικτες διαδικασίες και τίποτα δεν είναι απόλυτα παγιωμένο. Μπορούμε να εξετάσουμε και δυνατότητες μελλοντικής βελτίωσης της κατάστασης, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια δομή η οποία έχει προταθεί για την Όλαφ και πιστεύω ότι με τακτικές ανταλλαγές απόψεων σε σχέση με συγκεκριμένες πολιτικές για τα θέματα της καταπολέμησης απάτης και σε σχέση με το σχέδιο της μελλοντική εργασίας για την Όλαφ μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και το διάλογο κρατώντας πάντα μια διάκριση μεταξύ της συζήτησης για το ρόλο της ΟΛΑΦ και των συγκεκριμένων ερευνητικών και ανακριτικών δραστηριοτήτων της ΟΛΑΦ που πρέπει φυσικά να παραμείνουν απόλυτα ανεξάρτητες. Κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η σχέση της ΟΛΑΦ με τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο εμεί προτείναμε είναι να υπάρχουν τα σημεία αναφοράς τα σημεία επαφής στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο θα διευκολύνει την διάδραση της Όλαφ με τις εθνικές αρχές στα κράτη-μέλη. Είναι γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι τόσο πολύπλοκες οι δομές που ορισμένε φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να βρούμε ένα συνομιλητή, ένα θεσμό με, τον οποίο να μπορούμε να έχουμε τακτική επαφή από την πλευρά της Όλαφ. η δημιουργία <clears throat> σημείων αναφορά στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι φορεί. Απλώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν του αρμόδιου φορεί, οι οποίοι θα είναι κατά σημεία επαφή και αναφορά σε σχέση με την Όλαφ και θα δίνουν όλε τι απαραίτητε πληροφορίε και συμβουλέ προ την Όλαφ μέσα στα πλαίσια τη ερευνητική και ανακριτική εργασία. και επίσης σε σχέση με την ε, δικαστική συνέχεια των ερευνών της Όλαφ στο σχέδιο της πρότασής μας έχουμε περιλάβει και την απέτηση στα κράτη-μέλη να δίνουν τις δικές τους πληροφορίες στην Όλαφ για την κατάσταση της ε, δικαστικής συνέχειας που ενδεχομένως δίνεται σε μια έρευνα της Όλαφ. Εμείς προτείναμε όχι να γίνεται αυτό σε τακτά διαστήματα, αλλά να γίνεται αιτήση της Όλαφ ώστε να εξασφαλίσουμε και την μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στο σύστημα. Και για να μην δημιουργήσουμε ένα υπερβολικό διοικητικό άχθος για τα κράτη-μέλη. Είναι απαραίτητο όμως να υπάρχουν σαφείς διατάξεις στον κανονισμό που να προβλέπουν ότι όταν η Όλαφ ζητήσει από τα κράτη-μέλη τις ε, σχετικές πληροφορίες, τα κράτη-μέλη να είναι υποχρεωμένα να δώσουν όλες τις απαραίτητε πληροφορίες στην Όλαφ σε σχέση με τη δικαστική συνέχεια που δίδεται σε μια υπόθεση. Και να μπορεί επομένω η Όλαφ να αξιολογήσει το πώ προχωράει αυτή η διαδικασία σε δικαστικό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα το διορισμό του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ, Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με την διαδικασία διορισμού, η τελευταία διαδικασία που έλαβε χώρα προχώρησε με τρόπο πάρα πολύ ομαλό. Αυτό καταδεικνύει ότι έχουμε μια καλή σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Συγγνώμη, μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε και τις νομοθετικές ρυθμίσεις και πρόνοιες ότι δηλαδή η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο προτού κάνει τις προτάσεις για, την, για το διορισμό ενός νέου Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση του Συμβουλίου και η θέση του Κοινοβουλίου προτού γίνει η τελική απόφαση Κομισιόν για την πρότασή της. <clears throat> Αυτό έλαβε χώρα. Όταν έγινε ο διασμός του Τζοβάνι Κέσλερ ως ε, Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας επίσης και το γεγονός ότι η ΟΛΑΦ είναι μια υπηρεσία η οποία εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο τελικός διορισμός του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να γίνει από την ίδια την Κομισιόν, αλλά με πλήρη σεβασμό των θέσεων που θα έχουν διατυπώσει και το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο. το δεκαθεστώς της ε, Όλαφ η ύπαρξη ενός γενικού διευθυντή ο οποίος είναι αρμόδιος για την Όλαφ περιορίζει και τις δυνατότητες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λόγω του γεγονότος ότι η Όλαφ περιλαμβάνεται στην εσωτερική δομή της Κομισιόν. Υπάρχουν περαιτέρω τα θέματα που έχουν να κάνουν με, με το επιχειρησιακό εγχειρίδιο της Όλαφ. Έχουμε ένα τέτοιο εγχειρίδιο, το οποίο είναι δημοσιευμένο και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Όλαφ. <clears throat> Επομένως είναι προσβάσιμο σε όλους, έχει πλήρη, χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια. Όλα τα δικονομικά δικαιώματα και διασφαλίσεις που αναφέρονται εδώ πέρα στο τροποποιημένο νομοθετικό έγγραφο της Κομισιόν θα αντανακλώνται και, στην, ε, και στο εγχειρίδιο αυτό <clears throat> και το οποίο επομένω θα διατηρήσει απόλυτη διαφάνεια και θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων και οι κοινοβουλευτικοί. Αυτό λοιπόν θέλω να τονίσω σε σχέση με το εγχειρίδιο και το εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρόνοιες για την προστασία των εμπλεκομένων και θα δίνει σαφείς κανόνες ε, συμπεριφοράς για τους ερευνητές της όλα. Και όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σε σχέση τώρα με τις ε, τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποιες ενεκρίτησαν και ποιες δεν ενεκρίτησαν. Έχουμε ένα πίνακα που έχουμε προετοιμάσει και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να σας διαβιβάσω αυτά τα στοιχεία, να σας δώσω τον πίνακα τον αντίστοιχο στα μέλη του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορείτε κι εσείς να δείτε ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία πριτάνευσαν για να γίνει δεκτή ή όχι μια τροπολογία ιδίως στις περιπτώσεις που δεν, δεν είναι δεκτή μια πρόταση του Κοινοβουλίου. Αυτά που είπε ο Μπαρτ χάρη για την προστασία των δημοσιογράφων, των δημοσιογραφικών πηγών. Αυτή η προστασία προβλέπεται σε άλλα νομοθετήματα και οι νομομαθείς της Κομισιόν ανέφεραν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για να υπάρξει μια ειδική μνήα της προστασίας των δημοσιογραφικών πηγών στην νομοθεσία της ΟΛΑΦ. Καλύπτεται λοιπόν από άλλα νομοθετήματα αυτή η προστασία των δημοσιογράφων. Και σε άλλα σημεία μπορούμε να σας δώσουμε αυτό το συγκριτικό πίνακα για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου και προφανώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός <clears throat> ότι η πρόταση του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε και στο έγγραφο αυτό προβληματισμού το οποίο παρουσιάστηκε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το έγγραφο αυτό προβληματισμού και η αναθεωρημένη μας πρόταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απόψεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου και ως φορές αυτές οι θέσεις <clears throat> είναι αντίμαχες, δεν είναι πάντα σύμφωνες. Και ο στόχος της Κομισιόν φυσικά είναι να προσπαθήσει να εξεύρει μια συμβαστική λύση μεταξύ των δύο θέσεων για να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση η οποία μπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Σε σχέση τώρα με τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Εδώ η ιδέα της Κομισιόν ήταν πάρα πολύ απλή. Να έχουμε μια θητεία η οποία δεν ανανεώνεται γιατί η μη ανανεωσιμότητα δίδει περαιτέρω διαφυλάξει σε σχέση με την ανεξαρτησία του διευθυντή της, του Γενικού Διευθυντή Όλαφ. Στο τέλος της θητείας του λοιπόν δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι είναι αρμόδιοι για, την, για το διορισμό του ή τον επαναδιορισμό του, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της θητείας του τελείωσε. Δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα ανανέωσης της θητείας σου. Υπάρχουν βέβαια εδώ διαφορετικά συστήματα για, την, ε, για το διορισμό ανεξαρτήτων γενικών διευθυντών και ανεξαρτήτων αρχών και φορέων από την εμπειρία όμως που εμείς έχουμε συσσωρεύσει και από αυτά που έχουμε δει σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρούμε ότι μια πρόταση μη ανανεώσιμη θητείας είναι η πιο επωφελής για να εξασφαλιστούν τα θέματα της ανεξαρτησίας του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Και τέθηκε από την κυρία Αντρίεσεν ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τον αριθμό των μελών του προσωπικού στον τομέα του, των διαφορετικών ταμείων. Ίσως ο κύριος Κέσλερ θα μπορούσε εδώ να μας απαντήσει γιατί θα έχει περισσότερα στοιχεία. Είναι αυτός ο οποίος είναι αρμόδιος, αποκλειστικά μάλιστα αρμόδιος ως Γενικός Διευθυντής της ΟΛΑΦ για τα θέματα του προσωπικού και εγώ ως Επίτροπος δεν μπορώ να παρέμβω στις δραστηριότητες του. Και θα ζητήσω λοιπόν από τον Τζοβάνι να δώσει μία απάντηση στο ερώτημα αυτό. Αν έχει να πει κάτι. Επίσης μπορεί να προσθέσει και για άλλα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής θέλω να χαιρετήσω τον ε, Γενικό Διευθυντή, τον Τζοβάνι Κέσλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάω Ιταλικά, μιλάω Ιταλικά, ναι. Για την ερώτηση της κυρίας Ανδρεάσεν, εγώ δεν γνωρίζω να, έχουν μειωθεί, να έχει μειωθεί ο αριθμός των ελεγκτών σε καμία από τις υπηρεσίες μου, τουλάχιστον από την ε, άφηξή μου και μετά. Και παρόλο που ήρθα σχετικά πρόσφατα αυξήθηκε ο αριθμός των ελεγκτών. Αφαιρέθηκε ένας υπάλληλος από τους συμβούλους του Γενικού Διευθυντή και έγινε ελεγκτής. Επίσης, μέσα στην Όλαφ ξεκινήσαμε μία διαδικασία internal review procedure, μία εσωτερική αναθεώρηση των εσωτερικών μας διαδικασιών, δηλαδή του εγχειριδίου, του τρόπου με τον οποίο οργανώνουμε τις, τους ελέγχους, <coughs> κατά τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να τις απλουστέψουμε και να τις επιταχύνουμε. Αλλά επίσης, και κατά τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το δυναμικό που έχουμε στο, στα γραφεία μας, για να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια και προσωπικό ελεγκτικές δραστηριότητες αλλά και να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε καλύτερα και αυτό να φαίνεται δηλαδή και στο οργανόγραμμα στους δύο βασικούς μας στόχους δηλαδή τον έλεγχο κατά των απατών και την πρόληψη των απατών policy making δηλαδή εμείς έχουμε σαφώς υπόψη μας ε, στις αλλαγές που κάνουμε και θα κάνουμε στους επόμενους μήνες την μεταρρύθμιση, την αλλαγή ε, για να είμαστε έτοιμοι όταν θα εγκριθεί. Και αν μπορώ πρόεδρε, μια που έχω το λόγο, να πω και δύο γενικότερα πράγματα για την ε, πρόταση τροποποίησης του κανονισμού που μετά από τόσα χρόνια πρόκειται για μία αλλαγή υποχρεωτική θα έλεγα για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και σε μία ε, νομολογία που ήδη έχει δημιουργηθεί. Η Όλαφ έχει εμπλακεί στην διπηρεσιακή διαβούλευση της Κομισιόν και είχε και την πρωτοκαθεδρία σε όλη αυτή την διαδικασία και είχαμε την δυνατότητα να πούμε τη γνώμη μας και όσο με αφορά εμένα ε, ως ε, νέος γενικός διευθυντής ήρθα την τελευταία στιγμή. Αλλά η Επιτροπή και ο Επίτροπος μου έδωσαν την δυνατότητα, διακόπτοντας όλη την διαδικασία για μία περίοδο, μου έδωσαν τη δυνατότητα να εξετάσω το κείμενο το οποίο συζητεί το μέσα στην Κομισιόν και αφού διαβουλεύθηκα με τους διευθυντές μου διαπιστώσαμε 12 σημεία τροποποίησης του κειμένου που κυκλοφορούσε εσωτερικά και 11 από αυτά τα σημεία εγκρίθηκαν και βρίσκεται βρίσκονται στο εκτός από ένα δηλαδή και βρίσκονται στο κείμενο το οποίο σας προτείνεται σήμερα. Αυτό το κείμενο μπορεί να συμπληρωθεί. Εγώ από μια πλευρά θα έλεγα ότι το θεωρώ ακόμα ιδιαίτερα ρυθμιστικό, μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες, διότι ο καθένας έχει την απέτηση και το κοινοβούλιο φυσικά θέλει να, θέλει να προσθέσουν ένα κομμάτι, ένα ρυθμιστικό κομμάτι. Πρέπει όμως να καταβληθεί μια προσπάθεια για να δούμε κατά πόσο αυτοί οι κανόνες είναι συμβατοί. Δηλαδή από τη μια λέμε για παράδειγμα να κάνουμε γρήγορους ελέγχους αλλά από την άλλη μεριά επιβάλλουμε ε, ένα σωρό άλλες ε, ε, πρακτικές που τείνουν να καθυστερούν τις έρευνες. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για ένα καλό κείμενο. Και τόσο εγώ όσο και οι Όλαφ είμαστε στη διάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να σας βοηθήσουμε για να δούμε σημείο προς σημείο τους όρους αυτής της ρύθμισης. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ για την παρουσίασή τους και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Καλδέιρα Σίλβα. Πρόεδρε, ένα σημείο γρήγορα έχει προβλεφθεί να έρθει ο κύριος Κέσλερ εδώ σε αυτή την επιτροπή για να μας παρουσιάσει το σχέδιό του για την Όλαφ όπως μας αναφέρθηκε σήμερα το πρωί κατά την συνεδρίαση με την Επιτροπή Εποπτείας. Ναι, ναι, λέει ο Πρόεδρος, σύμφωνη λέει η κυρία Γιάλα. Καλησπέρα Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Αυτή η ακρόαση έπεται της ακρόασης του κυρίου Ενίρδα, ο οποίος ε, είχε, κάνει, είχε προβεί σε δηλώσεις στον Ολλανδικό τύπο. Τον ακούσαμε λοιπόν αυτόν τον κύριο εχθές στην Επιτροπή μας και πριν προχωρήσουμε σας το λέω ότι αναμεταδίδεται δορυφορικά η συνεδρίασή μας. Ο κύριος Καλδέιρα μου είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση καταρχήν αλλά είναι έτοιμος να ακούσει κατευθείαν τις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών και στο τέλος θα κάνει μια σύντομη συμπερασματική δήλωση. Ο κύριος Στάις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καλδέρα, σας ευχαριστώ που ήρθατε για να μας αναφέρετε την τις δηλώσεις ε, του κυρίου Εγγέντα στο Volksgrand ε, τον Δεκέμβριο που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί μακρόν μαζί του εχθές. Αυτό το οποίο θέλω να ξέρω είναι το εξής. Όταν είχατε... Όταν ήρθε στα χέρια σας αυτή η συνέντευξη μεταφρασμένη την πρώτη φορά, τι σκεφτήκατε, αναγνωρίσατε το θεσμικό σας όργανο σε αυτήν τη συνέντευξη ή σκεφτήκατε αυθόρμητα ότι σας φαίνεται κάτι το σουρεαλιστικό. Άλλη ερώτηση. Μερικές μέρες μετά από την συνέντευξη ο κύριος Ελγκβίρντα έστειλε μία επιστολή στην Volkskrant με διορθώσεις όπου ανακαλούσε μερικά από τα λεγόμενά του. Αυτό το οποίο μας εξέπληξε ήταν πόσο ο κύριος Εγκβίρντα έφτρασε τόσο γρήγορα, ε, τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα και έστειλε τη διορθωτική επιστολή, διότι συνένεσε στην δημοσίευση αυτής της συνέντευξης. Ο κύριος Εγκβίρντα διάβασε το σκρίπτ αυτής της συνέντευξης και έξι μέρες μετά ανακαλεί αυτό πραγματικά μας μπέρδεψε. Γιατί κατά τη γνώμη σας ασκήθηκαν πιέσεις, εξωτερικές πιέσεις στον κύριο Εγκβίρδα. Οι πρώην του συνάδελφοι του άσκησαν πιέσεις, ναι ή όχι. Το ελεγκτικό συνέδριο ή εσείς ο ίδιος ως πρόεδρος ασκήσατε πιέσεις κατά του κυρίου Εγκβίρντα. Υπάρχουν ε, τρόποι ε, ούτως ώστε ο κύριος ε, Εγκβίρντα να αναγκαστεί να ανακαλέσει τις δηλώσεις του ή να τις αλλάξει διότι μας είπε ότι μετά από πολλά χρόνια συμμετοχή στο ελεγκτικό συνέδριο διοντολογικά υπήρχαν δυσκολίες. Ασκήθηκαν πιέσεις από τα έξω και μετά από την δημοσίευση τη συνέντευξη συναντήσατε τον κύριο Εγκβίρντα, ναι ή όχι. Παρακαλώ πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Στράσκη για τα ερωτήματά του. Όταν έφτασα στο 2000 στο ελεκτικό συνέδριο, ήταν ένας διαφορετικός θεσμός ήδη από ό,τι είναι τώρα. Επομένως, όταν είπα ότι έχει, κάνει, έχει διατρέξει μακρό δρόμο το ελεκτικό συνέδριο τα 35 χρόνια της ύπαρξής του, αυτό νομίζω ότι αληθεύει, είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, σήμερα το θεσμικό μας όργανο είναι ένα αναγνωρισμένο, ε, ένας αναγνωρισμένος υψηλής ποιότητος φορέας που την χάνει γενικού σεβασμού. Και όπως είπα στα μέλη της Επιτροπής σας, η έκθεσή μας, εάν πρέπει να βαθμολογηθεί μεταξύ του 1 και του 4, έχει πάρει ένα βαθμό 3 τώρα. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βοήθησα ιδιαίτερα στην εξέλιξη αυτού του θεσμού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και μπορεί να εκδίδει εκθέσεις υψηλού επίπεδου. Όλα τα μέλη του θεσμού μας λοιπόν έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία. Χρειάζεται να τροποποιήσουμε να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον λογιστικών ελέγχων. Πριν από 35 χρόνια ήταν τελείω διαφορετική η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι είναι σήμερα, με έξι μόνο κράτη-μέλη. Τώρα είναι 27. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ασύγκριτα διαφορετικός από αυτό που έχουμε σήμερα. Έχει λοιπόν ε, εξελιχθεί τα πράγματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει, νέες, έχει αποκτήσει νέες αρμοδιότητες και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο επίσης. Αυτά που είπε και ο Σενκβίντ είναι κατά κάποιο τρόπο τα απομνημονεύματά του και οι αναφορές του ιστορικές σε ένα θεσμικό όργανο το οποίο κατάφερε να κερδίσει τη θέση ως ένα θεσμικό όργανο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταφέρεται και η σαφής κατεύθυνση την οποία έχουμε ακολουθήσει. Εδώ το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να ατενίσουμε το μέλλον για να δούμε πού είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι τα σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το θεσμικό μας όργανο βέβαια εποφελήθηκε και από τις ε, συμβολές του κυρίου Ένβιντα τα τελευταία χρόνια. Με τις εσωτερικές μας μεταρρυθμίσεις έχουμε καταφέρει να καλύψουμε όλες τις συστάσεις της, ε, του, του ελέγχου κατά κάποιο τρόπο των ομοτήμων και των προτάσεων των ομοτήμων. Και η Επιτροπή σας έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση και τις, ε, την εφαρμογή των προτάσεων των νομοτήμων. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουν όλοι ότι είμαστε ένας ανεξάρτητος φορέας, το ελεκτικό συνέδριο. Με ρωτήσατε επίσης αν εγώ ή κάποιος άλλος είχε ασκήσει πίεση στον κύριο Ενβίδα να αποσύρει τις ε, δηλώσεις του. Μα βέβαια και όχι. Ο κύριος Έγκβιδα πρέπει να υπομειστεί την πλήρη ευθύνη των λόγων του και των δηλώσεών του. Και χθες μπορέσαμε να το ρωτήσουμε αν έχει θεωρήσει ότι υπευλήθη σε πίεση από κάποιους. Εγώ του ανέφερα ότι δεν συμμεζόμαστε την άποψη που εξέφρασε στην συνέντευξή του, αλλά για τα λόγια του αυτός θα πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη και εξάλλου την απόλυτη ευθύνη για όλες τις δηλώσεις που έκανε μετά δημόσια σε διάφορες εφημερίδες με δική του πρωτοβουλία. Στο European Voice και σε άλλα μέσα όλα αυτά ήταν με την πρωτοβουλία του κυρίου του Εγκριντά. Δεν νομίζω ότι κάθε από αυτά είναι καινούργια. Ο κύριος έχει αναφερθεί άμεσα και στο προσωπικό του ελεκτικού συνεδρίου εξηγώντας τι εννοούσε και τι δεν εννοούσε. Κανείς δεν του το απίτησε αυτό, αλλά το έπραξε διότι θεώρησε ότι αυτό ήταν απαραίτητο για να υπάρχει σαφήνεια από την πλευρά των ελεκτών, που είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το όργανο όμως αυτό που είναι σήμερα. Η κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Καρδέιρα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Για να ξεκαθαρίσουμε αυτά που μας είπε και ο κύριος ε, Εγκβίρδα εχθές. Ε, που αναγνωρίσε το λάθος των δηλώσεών του, πώς τις παραποίησε ο τύπος ε, και μετά τις αναθεώρησε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λοιπόν στο ότι του ασκήθηκε πίεση κτλ. Σήμερα το πρωί με το ψήφισμα που εγκρίναμε αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε για το πώς θα διαχειριστούμε το μέλλον τα προβλήματα που διαμορφώνονται σε ένα τόσο πολύπλοκο θεσμικό όργανο που αυτοί που εργάζονται εκεί υπόκεινται σε στρες και πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να δώσουν και τον καλύτερό τους σε αυτό. Σας ευχαριστώ για την καλή σας διάθεση και σύμφωνα με το ψήφισμα που εγκρίναμε σήμερα το πρωί και που θα επικυρώσει ελπίζω η Ολομέλεια μπορούμε να διατηρήσουμε την συζήτηση για να βελτιώσουμε τη σχέση του Κοινοβουλίου, αυτής μας της Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνοδρίου. Και χαίρομαι που ο κύριος Εγκβίρ αναγνώρισε τη δική σας ε, περίοδο προεδρίας ως την πιο γόνιμη και την πιο καρποφόρα. Ελπίζουμε λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια του διαλόγου θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για τη βελτίωση όλων των θεσμικών οργάνων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σταθερά με το Κοινοβούλιο. Και θέλω να επιβεβαιώσω και πάλι όπως το έκανα πριν από ένα μήνα όταν παρουσίασα το πρόγραμμα εργασία μας στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή σας, ότι έχουμε μια ειδική σχέση με αυτή την Επιτροπή. Τα τελευταία 35 χρόνια το ελεκτικό συνέδριο έχει βασιστεί σε αυτή τη σχέση. Και θυμόμαστε τα πρώτα μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, τον κύριο Άικνερ, ο οποίο ήταν ο πρώτο πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Αυτή η στενή σχέση λοιπόν με την Επιτροπή σα, ο ρόλο που παίζει το Ελεκτικό Συνέδριο στη διαδικασία απαλλαγή, οι κοινοί στόχοι που συμμεριζόμαστε με την Επιτροπή σα, δηλαδή το να μπορούμε να ελέγχουμε αυτού που είναι υπόλογοι και να βελτιώσουμε την οικονομική διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθήσουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, να εντοπίσουμε τους κύριους χώρους όπου μπορεί να προκύψει μια βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και πιστεύω βαθύτατα ότι η νέα συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει δυνατότητες να οικοδομήσουμε από κοινού. Έχουμε νέους μηχανισμούς λογοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει η μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών προοπτικών. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν σημαντικές συνέπειες και απόρριες για την Επιτροπή σας και, την, και το Ελεκτικό Συνέδριο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και έχουμε επίσης πολλά να πράξουμε από κοινού για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των ευκαιριών που μας δίνει ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός. για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το σωστό έλεγχο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει και η χρηστή ε, λειτουργία του προϋπολογισμού. Επίσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τους νέους εποπτικούς φόρους για τις χρηματαγορές, για τις ασφάλειες και τα τραπεζικά ιδρύματα Έχουμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον, όπου και πάλι θα πρέπει να δούμε τον κατάλληλο τρόπο να καταλήξουμε σε μια σωστή διαδικασία λογιστικού ελέγχου. Και όπως σας είπα προηγουμένω, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία έναντι του <clears throat> απλού πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωση για όλα τα εργαλεία, είτε είναι χαρακτήρα διακυβερνητικού χαρακτήρα, και διαχειριστικού χαρακτήρα και των άλλων φορέων που είναι υποσυζήτηση τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουμε με ένα αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και από τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και περισσότερο για το πόσο διαφανής και υπόλογος είναι αυτός ο μηχανισμός και πόσο αξιόπιστα είναι τα στοιχεία επί των οποίων εδράζεται η λήψη αποφάσεων από αυτό το φορέα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας συγκεκριμένα μαζί με το Ελεκτικό Συνέδριο θα πρέπει να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι αυτή η διαφάνεια και η λογοδοσία προς το κοινό θα υπάρχει και θα υπάρχει και βελτίωση της ε, οικονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι από τους οποίους είναι εξάλλου κοινή μας ε, στόχη. Κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Καλντέρα. Εχθές κατέξτε πολύ τα σαφές από τον κύριο Μάτ τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Υπάρχει μια ε, προσπάθεια, την οποία ενισχύουν κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπορούσε και την ε, προβάλλουν προκειμένου να προκαλέσουν ε, αίσθηση στην κοινή γνώμη. Εγώ όμως θα ήθελα να συστήσουμε λίγο περισσότερο την ουσία, τα ζητήματα και την αλήθεια και σε ποιο βαθμό άσκησε το ελεγκτικό συνέδριο πίεση των μάτων προκειμένου να διορθώσει τις δηλώσεις του. Τι είδους συζητήσει λοιπόν έλαβαν χώρα. Διότι πιστεύω ότι χωρίς να είναι σκόπιμο αυτό ότι αυτή η συνέντευξη αποτέλεσε λίγο πολύ το μοχλό για την προαγωγή της μεταρρύθμισης του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχει προχωρήσει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση και ίσως ήταν πρόημη η προβολή στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πάντως για την ε, διάθεση να συζητήσουμε το θέμα αυτό, για την ε, πρόθεσή σας να μην συγκαλύψετε, να τρέψετε τη συγκάλυψη υπόθεση, αλλά αντίθετος να την αντιμετωπίσετε εγκαίρως. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν ε, περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Μάτεν ε, και εσύ είναι ακόμη ήδη στη σύνταξη, να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Και δεν θέλω να εξηγήσω γιατί, γιατί το συζήτησα και χτες αυτό. Υπάρχουν κάποιοι στο ελεγκτικό συνέδριο, οι οποίοι δεν θεωρούνται και τόσο επιτυχείς. Εάν, παραδείγματι, δούμε τις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές, οι ελεγκτικές αρχές καλύτερα, έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και μπορούμε να πούμε ότι στην, ε, στις εκθέσεις γενικά είχε πρωτοκαθεδρία στις προσπάθειες ε, για την ε, εξέταση των λογαριασμών. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος με πολλή εμπειρία και θα έλεγα, θα ρωτούσα λοιπόν να είστε διατεθειμένοι να τον αξιοποιήσετε, έστω και να έχει ήδη στοξιδοτηθεί. Thank you for your kind comments. Σας ευχαριστώ για τα τόσο καλά σας και αγαθά σχόλια. Αυτό είναι ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο συζήτηση μέσα στο ελεκτικό συνέδριο. Πώ να εκμεταλλευτούμε τα πρώην μέλη μας, όχι μόνο τον κύριο Εγκβιρντά, αλλά όλους αυτούς οι οποίοι υπηρέτησαν στο το ελεκτικό συνέδριο και μπορούν να μας δώσουν την εμπειρία τους και μπορούν να συμβάλλουν εποφελώς όχι μόνο στο σημείο αυτό που αναφέρατε για την μεταρρύθμιση του ελεκτικού συνεδρίου αλλά και για οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου η εμπειρογνωμοσύνη τους και η εμπειρία τους μπορούν να είναι πολύτιμες για μας. Το σκεφτόμαστε και είμαστε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε στο άμεσο μέλλον αυτές τις δυνατότητες. Αλλά πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Το ελεκτικό συνέδριο είναι ένας θεσμός. Τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου διορίζονται μέσω μιας σαφούς και αυστηράς διαδικασίας. Θα πρέπει να σέβονται το περιεχόμενο των συζητικών και το να, είναι κανείς, να έχει κάνει την ιδιότητα ενός πρώην μέλους του ελεκτικού συνεδρίου σημαίνει ότι μπορεί να δίδει συμβουλές, μπορεί να του ζητηθεί να δώσει τη γνώμη του για ένα έγγραφο και αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Δεν το έχω συζητήσει με τους συναδέλφους μου. Ίσως θα μου λέγανε ότι αυτά που λέω σήμερα δεν πρέπει να τα πω. Αλλά εγώ προσωπικά είμαι πολύ θετικός αν μπορώ να κλείσω τη θητεία μου με, την, ε, ε τα εγγένεια του νέου κτηρίου του Ελεκτικού Συνεδρίου, αν μπορώ να προσκαλέσω τα διάφορα πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου που θα μπορούσαν να συμβάλλουν με διάφορους τρόπους, θα ήταν πολύ θετικό για μένα. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι και το θέμα της έρευνας. Όπως ξέρετε το ελεκτικό συνέδριο ξεκίνησε ένα βραβείο ερευνητικό για καινοτομίες στον τομέα της, του λογιστικού ελέγχου και της λογοδοσίας και είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε περισσότερο αυτή την ιδέα. Θεωρούμε ότι οι πρώην μέλη του ελεκτικού συνεδρίου μπορούν να δώσουν μια πρώτη συμβολή ώστε να μπορέσει να προωθηθεί το θεσμικό όργανο στο οποίο όλοι με μεγάλη χαρά είμαστε μέλη. Ο κ. Γκαρμπέντη, σας ευχαριστώ. Και Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Καρδέλα που ήρθε και μας μίλησε με τόση ειλικρίνεια. Εξυπλάκη διαβάζοντα τελευταία συνέντευξη του κυρίου Έγκερντα. Είχα βέβαια και άλλε παλαιότερα, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είχαν τόσο πολύ διωγγωθεί από τα μέσα μα και ενημέρωση. Και έτσι πρέπει να πω ότι δεν εξεπλάγει τόσο από το περιεχόμενο, γιατί για το παρελθόν μιλούσε. Πλην όμω, θα ήθελα να πω ότι έχω τα εξή δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με πιθανέ ε, πιέσει πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι εμπειρία έχετε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στα σχέδια των εκθέσεών σας. Βεβαίως μπορείτε να δώσετε πιο πολλές ε, πληροφορίες να σας καλέσω να δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά οι πιέσει σε πιο βαθμό φτάνουν. Και επιπλέον τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου που θα ήθελα να επανέλθουν για μια δεύτερη και τρίτη θητεία. Και δεδομένου τα κράτη-μέλη έχουν λόγο στην ε, ανανέωση της θητείας. Κάποιος λοιπόν, ε, κάποιο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου ενδέχεται μήπως να είναι, πιο, να είναι λιγότερο επικριτικό έναντι του οικίου κράτους μέλους προκειμένου να κερδίσει την ανανέωση της θητείας του. Δεν θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθεί κανείς ε, πώς ε, πρέπει να λειτουργεί το ελεγκτικό συνέδριο και η έλεγχη, η διαδικασία του ελέγχου. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι ένα ε, όργανο με επαγγελματισμό που ασκεί με τρόπο επαγγελματικό την ελεγκτική του δραστηριότητα και ότι είναι σχεδιασμένο, ε, η οι, οι τρόποι σύνταξης μιας εκθέσεως ώστε να εξασφαλίσει αντικειμενικότητα και ουδετερότητα προφανώς δεν ε, έχει θέσει καμία συζήτηση ή αμφισβήτηση περί αντικειμενικότητας ή ε, ερώτηση περί πιέσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο ερώτημα βέβαια είναι τι θέματα προσδιορίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο προσδιορίζει με τις δικές του προδιαγραφές το αντικείμενο των ελέγχων του με τους στόχους που ορίζει το ίδιο και αυτό σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές τις οποίες με πολύ μεγάλη ευσέβεια τηρούμε. Βεβαίως, ταυτόχρονα κάνουμε και την επιτόπου έρευνα στην Επιτροπή, τα κρατημέλη, χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ε, εισπράττουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συλλέγονται λοιπόν στοιχεία με τις αυτοψίες αυτές, αξιολογούμε στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά, φροντίζουμε να τα επιβεβαιώσουμε και τα περνούμε σε μια διαδικασία λεγόμενη καθάρισης που είναι κατά τιμολίαν όπως θα γνωρίζετε ασφαλώς ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελεγχόμενο όργανο ή το κοινοβούλιο, είναι το κοινοβούλιο το ελεγχόμενο όργανο αυτό που λέμε κατά τιμολίαν διαδικασία. Και το ελεγχόμενο όργανο βέβαια έχει το δικαίωμα να δώσει απάντηση στις παρατήρησεις του λακτικού Συνεδρίου στη διαδικασία αυτή διευκρινίσως ή επιβεβαιώσεως των ε, ε, πορισμάτων μπορεί ασφαλώς να εμφανιστεί απόκληση απόψεων, μπορεί να γίνουν σημαντικές συζητήσεις. Ναι, αλλά το μόνο όργανο το οποίο μπορεί να αποφασίσει τι θα συμπεριλάβει στην έκθεσή του είναι το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο έχει τη μορφή ενός δικαστηρίου στο οποίο συμμετέχουν μέλη από ε, διάφορα κράτη-μέλη, πέντε το καθένα, με την ε, ε, συλλογική μορφή, όπου δηλαδή το κάθε μέλος στην κάθε επιτροπή που συμμετέχει μπορεί να έχει διαφορετική άποψη και να την εκφράζει, αλλά άπαξ και εκδοθεί η άποψη, είναι, η γνώμη είναι δεσμευτική για το σύνολο του οργάνου. Και ως εκ τούτου, η αδίποτε παρέμβαση, η προσπάθεια επιρροής από, κάποιον, από κάποιο μέλος που ενδεχομένω ενδιαφέρεται για την ανανέωση της θητείας του με την υπόνοια ότι μπορεί να συμπεριφέρεται κατά τρόπο διαφορετικό ε, για να εξασφαλίσει την ε, επανεκλογή του από το γεγονός και μόνο ότι έχουμε αυτή την συλλογική μορφή, δηλαδή την ε, ε, λειτουργία ως σύνολο, δεν μπορεί να επηρεαστεί το ελεκτικό συνέδριο από ένα μέλος ή από μια κυβέρνηση. Και η εμπειρία που έχουμε Ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον από το 2000 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έχω ο ίδιος περάσει την ανανέωση της θητείας αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έκανα ήταν όταν το, το Συμβούλιο ενημέρωσε το κράτος μέλος μου ότι θα λήξει η θητεία μου ήταν να απευθυνθώ στο κράτος μέλος, να μίλησω με τον ε, αρμόδιο υπουργό και να πω είμαι στη διάθεσή σας. Ε, λίγη θητεία μου την τάδε ημερομηνία και πολύ ευχαρίστω να ξαναπροσφέρω για τα επόμενα έξι χρόνια τι υπηρεσίε μου στην πατρίδα μου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά την απόφαση θα τη εσεί. Πιστεύω λοιπόν ότι την ίδια κίνηση έχουν κάνει όλοι οι συναδελφοί μου. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι το γεγονός πως η διαδικασία περνάει από μια διαδικασία διορισμού από τα κράτη-μέλη η ανανέωση της θητείας μπορεί να επηρεάζει την αντικειμενικότητα ή την ανεξαρτησία των μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό όμως ότι είναι σαφές. Η διαδικασία που ισχύει εξασφαλίζει ανεξάρτητη ελεγκτική δράση με την έκθεσή μας και περιέχει πολλές διασφαλιστικές λικλίδες ώστε να μην ε, μπορεί κανείς να ασκήσει πίεση στα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου, για οδήποτε λόγο ή υπό οποιοδήποτε όρο. Γιατί πέραν των άλλων έχουμε και σαφείς διαδικασίες για να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα είναι όλες οι ελεγκτικές μας δράσεις ε, αντικειμενικές και ουδέτερες. Είναι, είναι αδύνατο δυνάμει των διαδικασιών που ισχύουν αυτή τη στιγμή να εντοπίσετε κάποια περίπτωση, να βρείτε κάποια περίπτωση επιρροής ή παρέμβασης όπως την επενεχθήκατε. Είναι 100% ασφαλής η διαδικασία. Στεγανή 100%. Και πιστεύω ότι εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε εμπιστοσύνη στο ελεγκτικό συνέδριο, πρέπει αυτό να το καταστήσουμε απολύτως σαφές. Πιο σαφές λοιπόν ουσιαστικά θα ήταν να μην υπάρχει υπενιγμός περί ε, επιρροής επειδή ενδεχομένως ε, υπάρχει η διαδικασία της ανανέωσης αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί στην ε, διαδικασία των θεσμικών οργάνων. Δεν οφείλεται μόνο δηλαδή στην ανανέωση της εντολής, στην πιθανότητα ανανέωση της εντολής είναι κάτι που ισχύει για όλα τα όργανα, όχι μόνο το ελεγκτικό συνέδριο, για κάθε όργανο, γιατί αν θα πρέπει η θητεία του να είναι πιο μακρά, πιο σύντομη, αν πρέπει να είναι ανανεώσιμη ή μη. Ασφαλώς, πολλές διαφορετικές επόψεις μπορεί να ε, υπάρχουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως έχουμε το, το δικαστήριο για να τα πω στα γαλλικά, είναι απόλυτα απόλυτα προστατευμένο, ανοσοποιημένο από τέτοιου είδους επιμολύνσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Στάς. Μια ερώτηση. Μια κύριε Πρόεδρε. Για τον κύριο, ε, σε σχέση με το είπε ο κύριος Κερμπράντε λέτε ότι, είστε, α, ότι έχετε ανοσία στις πιέσεις. Ο κύριος Εγκβιρντόρ μας είχε πει όμως στην ακρόαση του ότι το 2005 ο κύριος Κάλλας, αρμόδιος για την πάταξη της διαφθοράς επίτροπος, είχε παρέμβει. Είχε κάνει μια επέμβαση στο ελεκτικό συνέδριο είχε πει ο κύριο Σουτό ότι είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τη μεθοδολογία του ελεγκτικού συνεδρίου και μα λέτε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν ψέματα, δεν υπήρξε παρέμβαση του Επιτρόπου Κάλλα ούτε στο πρόσωπό σα ούτε στο πρόσωπο κάποιου άλλου ε, μέλου του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό είναι μια άμεση ερώτηση και απαιτείται άμεση απάντηση. Σα ευχαριστώ. Αν θυμάμαι καλά. Ήμουνα σε μια συνεδρία της Επιτροπής σας στο Στρασβούργο όταν παρουσιάστηκε, στην οποία παρουσιάστηκε μάλλον, η ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για εκείνη τη χρονιά. Και αυτό το οποίο, αν αναφέρεστε σε αυτά τα οποία ελεγχθεί σαν τον κύριο Κάλλας, ναι, υπήρξε πίεση βέβαια από την Κομισιόν, αλλά με έναν τρόπο απόλυτα διάφανο και ο κύριος Ενκ Βίντρα μάλλον αναφέρεται σε εκείνη την ε, χρονική στιγμή γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια άλλη στιγμή στην οποία αναφέρεται ο κύριος Ενκ Βίδρα. Κάθε θεσμικό όργανο όμως έχει μια διαφορετική άποψη για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κάθε θέμα. Εγώ χαίρομαι που βλέπω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει βρει το σωστό τρόπο για την ανάκτηση των κονδυλίων και τα θέματα της δημοσιονομικής διαφθοράς. Είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μια διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα του Ταμείου Συνοχής κτλ. Αν λοιπόν υπάρχει, υπήρξε πίεση, νομίζω ότι τελικά αυτή η πίεση οδήγησε σε μία από τις καλύτερες λύσεις για τα θέματα αυτά και η Κομισιόν ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εργασίας για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά Εγώ δεν ήμουν παρόν χθε, δεν, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Σέγγβίδρα ή τι δεν είπε. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι αν αναφέρθηκε ο κύριος Σέγγβίδρα σε αυτό που έγινε πριν από έξι χρόνια στο Στρασβούργο παρουσία του κυρίου Κάλλα. το κατανοώ, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ κάποια άλλη τέτοια ευκαιρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν δεν έχετε μια τελική δήλωση. Οι ερωτήσεις έχουν τελειώσει. Ε, I want to thank for Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το χρόνο που μου δώσατε και την ευκαιρία μου δώσατε να λάβω το λόγο ενώπιόν σας και χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι το ανεξάρτητο ελεγκτικό συνέδριο έχει παραμείνει ανεξάρτητο και έχει ενισχύσει τις πρωτοβουλίες του. Η συνθήκη δίνει στο ελεγκτικό συνέδριο μια σειρά από διαφυλάξεις που αφορούν το καθεστώ μας, καθεστώς μας ως θεσμό, τη διαδικασία διορισμού των μελών του ελεκτικού συνεδρίου και τον συλλογικό χαρακτήρα των αποφάσεών μας. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέλος μπορεί να συζητήσει μια έκθεση αλλά, του ηλεκτρικού συνεδρίου, αλλά μια έκθεση η οποία εγκρίνεται δεσμεύει όλα τα μέλη μας. Η αντικειμενικότητα των εκθέσεών μας και η αμεροληψία τους <clears throat> είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και από τους ομοτήμους μας. Η αναθεώρηση από ομοτήμους που έγινε το 2008 ήταν πολύ θετική από αυτή την άποψη. και κατέληξε στο ότι το Συμβούλιο έχει δημιουργήσει ένα σωστό πλαίσιο το οποίο καλύπτει τις διεθνείς πρακτικές. Ότι οι εκθέσεις μας βασίζονται σε στοιχεία τα οποία είναι ε, εδρεωμένα και ότι οι εμπλεκόμενοι έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις εκθέσεις μας. Αυτά τα συμπεράσματα έχουν επίσης επιβεβαιωθεί και στις επαφές με μέλη της Επιτροπής σας και με εμπλεκόμενους στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι ένα επαγγελματικό όργανο για λογιστικό έλεγχο το οποίο συνεργάζεται έντονα για την ανάπτυξη λογιστικών ελέγχων στο δημόσιο τομέα μέσω της συμμετοχής μας σε διεθνείς οργανισμούς εμείς βοηθούμε την ανάπτυξη των διεθνών προτύπων <clears throat> για λογιστικούς ελέγχους. Είμαστε επίσης ε, σε στενή επαφή με τις επιτροπές των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων και ε, αναπτύσσουμε κοινέ μεθόδους για τον έλεγχο των Ευρωπαϊκών Διαθροντικών Ταμείων. Και βοηθούμε αυτή τη στιγμή σε μία αναθεώρηση του ελεκτικού φορέα της Νορβηγίας. Όλα τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει για να επιτευχθεί να είναι το ελεκτικό συμβούλιο αυτό το οποίο είναι σήμερα. Εμείς έχουμε προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες στο περιβάλλον λογιστικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρόσφατες αλλαγές το έκαναν ικανότερο να αντιμετωπίσει και να προβλέψει τις μελλοντικές αλλαγές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ελεκτικό συνέδριο, όπως ξέρετε, έχει μια στρατηγική μεγιστοποίησης του αντικτύπου του αερού της και καλύτερης δυνατής χρήσης των πόρων του. Και έχουμε ε, αναθεωρήσει τις διαδικασίες διακυβέρνησής μας, έχουμε δημιουργήσει και ένα σύστημα με τμήματα για να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη λήψη αποφάσεων. Κύριε Πρόεδρε, τον εργαζόμαστε αποτελεσματικά με τους εμπλεκόμενους, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή σας κτλ. Όλα αυτά είναι κομβικά για την μελλοντική μας επιτυχία. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Κοινοβούλιο που βασίζεται στις ιστορικές μας σχέσεις, στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη και στην στενή σχέση που έχουμε με την Επιτροπή σας. Θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω και να ξαναυπογραμμίσω όλα αυτά τα θέματα κλείνοντας προσβλέπουμε στη συνέχιση της εργασίας μας μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινέ προκλήσεις για να βελτιώσουμε την οικονομική διαχείριση και την λογοδοσία και διαφάνεια προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. E Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό βράδυ. Σε αυτό Μία αυτό θα περάσουμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης πριν από την ε, συνεδρία των συγκομιστών. Απαλλαγή 2009, Γενικός Προϋπολογισμός, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Χατζημάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατέθεσαν πάνω από 100, 300, 304 τροπολογίες για την σχετική με την απαλλαγή. Θα ήθελα να σχολιάσω. Το αυτό το βιβλίο του πέκ, είναι ενδιαφέρον. Ορισμένα πράγματα και να ευχαριστήσω την Επιτροπή για μια δεύτερη επιστολή που μας, ε, μου απέστειλε. Την οποία πρόωθησα με διάφορα στοιχεία για να δοθούν απαντήσεις στους συναδέλφους. Διάφορα στοιχεία. Ευχαριστώ λοιπόν. Πάντως πιστεύω ότι ε, υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν ακόμη απαντήσεως σύντομα. Στο σημείο α έως σιγματάφ. Πρώτον, ε, διαχείριση. Στο α, ευχαριστούμε την Επιτροπή που μας ε, παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές οι δύο τροπολογίες των συναδέλφων σε ένα βαθμό ορισμένες μάλλον αποδυναμώνουν τις ε, θέσεις του εισηγητού, άλλες δε την, τις ενισχύουν. Ο εισηγητής λοιπόν εγώ θα πρότεινα και στον ε, κατάλογο των ψηφοφοριών οι συναδέλφοι να δεχθούν την μέση εδώ, την αρχική πρόταση δηλαδή. Και στο στάδιο αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να συνταχθούν συμβαστικέ τροπολογίε. λόγω της φύσεως αυτών των τροπολογιών. Δεν είναι εύκολο μερικές φορές να συνενωθούν σε ένα κείμενο. Για το συγκεκριμένο θέμα πάντως θα ήθελα να επισημάνω ότι καλό θα είναι να μην αποθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στο θέμα της απάντησης ε, των ε, προσδοκιών αυτών, σε ανταπόκρισεις προσδοκίες και να μην αποδυναμώσουμε το κείμενο. Για το Β ε, θέμα, δηλαδή για την υπογραφή του αρμόδιου επιτρόπου, θα ήθελα να επισημώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο ήταν πολύ συνεργάσιμη, αλλά ανταποκρίθηκε πάρα χρήμα. Και ζήτησε από όλους τους επιτρόπους μια σαφή ε, ενημέρωση και ανταλλαγή μεταξύ των γενικών διευθυντών που ουσιαστικά υπογράφουν αυτές τις ε, εκθέσεις δραστηριοτήτων και των ε, οικείων επιτρόπων. Η κυρία Ντέ, γενική γραμματέα της Επιτροπής το έπραξε. Τα κύρια στοιχεία λοιπόν, ίσως όχι επιτροπή, όχι η υπογραφή του επιτρόπου, αλλά η φύση, το πνεύμα ε, Αυτή τη συνεργασία και της ευθύνης ικανοποιούνται νομίζω. Ως εκ τούτου εγώ συμφωνώ σε κάποιες από τις τροπολογίες των συναδέλφων, τη 261 και την 263 ειδικότερα, μέχρι 266, του κυρίου Ιβάν και του κυρίου Μπέλντερ, πλήστορ. Τις δέχομαι και ως εκ τούτου, αν δεν τυπώνω το αρχικό μου κείμενο, για να ευθυγραμμιστεί περισσότερο στα όσα έχει αρχικά ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα έχει δώσει πολύ καλές απαντήσεις και ευχαριστώ τον κύριο Ιβάν και τους συναδέλφους. Το τρίτο τμήμα. διακοπή ή άρση των πληρωμών. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσέφερε πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές ή ε, άρσεις πληρωμών ε, στη δεύτερη επιστολή. Έχει δώσει τα στοιχεία αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με πληροφορίες που αφορούν και προηγούμενα έτη, το 2010. Πράγμα το οποίο κρίνουν προφανές. Βεβαίως είναι πιστός πληροφορίες να αφορούν το 2010 και το 2011 γιατί μόνο το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο, το μέσον της ε, διακοπής. Θα ήθελα ωστόσο και εγώ να αναφερθώ στο κείμενό μου στην αυτόματη διακοπή ε, και μια πρόταση να αντικατασταθεί αυτός ο όρος από τον όρο συστηματική διακοπή. Αυτό σε τελευταία ανάλυση είναι αυτό που πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όχι μόνο δίνει στοιχεία δημόσια ε, για τα κράτη-μέλη και μια διαδικασία διακοπή πληρωμών, αλλά ταυτόχρονα δίνει και κατευθυντήριε γραμμέ με πληροφορίε κατά τρόπο συστηματικό ή μέσα σε ένα σύστημα για το πότε πρέπει να λαμβάνει η χώρα αυτή η διακοπή της ε, καταβολή των ποσών. Και γι' αυτό ακολουθώ αυτή την διατύπωση του συναδελφού Ιβάνου από την τροπολογία του. Στην τροπολογία 269-270 συγκεκριμένα. Για τη 278 πάλι δική σας κυρία Ιφάν. Εγώ προτείνω, αντιπροτείνω μια προφορική τροπολογία για να προσαρμόσουμε το κείμενο στη γενικότερη δομή του εγγράφου μου. Το αυτόματι λοιπόν να το αντικαταστήσουμε με ένα συστηματική. Αυτό είναι μια προφορική τροπολογία, όπω είπα. Και επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Ακόμα περιμένω κάποια στοιχεία για προηγούμενα έτη, όπω μου το έχετε υποσχεθεί. Προχωρώ στο σημείο Δέλτα. Βελτίωση των διορθωτικών μηχανισμών. όπου Μέχρι τις παρούσες δεν έχουμε λάβει πληροφορίες. Από ό,τι φαίνεται είναι και το πιο ε, δύσκολο έργο για την Επιτροπή. Δηλαδή θα πρέπει να κάνετε αναδρομή σε προηγούμενα έτη και δεν είναι εύκολο να αναζητήσετε, να βρείτε τις λύσεις, τις απαντήσεις ε, και τις πληροφορίες. Αλλά αν πάση έχετε προσχεθεί ότι μέχρι τέλη Απριλίου θα έχουμε τα στοιχεία, εγκαίρως δηλαδή και πριν από την ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Και θα ήθελα να καλωσορίσω όχι μόνο τον κύριο Φλιέρνερ που έρχεται, αλλά και να τον ενημερώσω τη δική του τροπολογία που αφορά το έτος ε, για το οποίο γίνεται αναδρομή στην αποκάλυψη στοιχείων για διορθωτικούς μηχανισμούς για το 2004, το 2000, τελεία, 2000. Προφορική τροπολογία. Πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό η Επιτροπή. Άλλωστε έχει συμφωνήσει με τις διαπραγματεύσεις. Και ευχαριστώ τον κύριο Φιέλναρ για το απολογείο του. Για το σημείο F. Σίγμα δηλαδή τη νέα λογική δαπανών, βελτίωση των δαπανών, του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι δαπανέ. Είχαμε μια πρόταση του κύριο Φιέλνερ για διαγραφή ολόκληρη παραγράφου και τη σχετική απέτηση θα πρότεινα να μην διαγραφεί ολόκληρη αυτή η απέτηση. Γιατί, διότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφέρει πολύτιμη, πολύτιμη ενημέρωση για αυτό το στόχο και ειδικότερα πολύ συγκεκριμένες και σαφείς προτάσεις απλούστευσης. Δεν θα ήθελα να την αποθαρρύνω. Γι' αυτό δεν δέχομαι την τροπολογία αυτή, κύριε Φιέλνερ. Ευχαριστώ πάντως για την πρότασή σας. Και ίσως αν δείτε τις νέες και φρέσκες ε, προτάσεις για την απλούστευση, νομίζω ότι θα δείτε πως είναι πολύ ε, εύκολο να μειωθούν τα ε, κατόφλια να εισαχθούν νέοι και απλοί κανόνες στις διαδικασίες προκηρύξεων δημόσιων προμηθειών και ίσως πιστείτε να αποσύρετε την τροπολογία σας. Και να πάω στις άλλες τροπολογίες τώρα. Ιδίω στις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, όχι μονάχα η κυρία Γκρέσλε, αλλά κυρίως η κυρία Γκρέσλε έχει καταθέσει κάποιες προτάσεις σε σχέση με το προσωπικό και τους κανονισμούς που το διέχουν. Οι κανονισμοί για τους υπαλλήλους έχουν να κάνουν με δαπάνες. Αυτό είναι ένα στοιχείο της απαλλαγής προφανώς. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω κάποιες από τις οπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί και τις έχω συμπεριλάβει στην εκθεσή μου. Μόλον τούτο είναι γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή για τα ειδικά αυτά σημεία είναι η νομική επιτροπή και γι' αυτό κάποιες από αυτές τις τροπολογίες θα ήθελα να αναδιατυπωθούν κάποιες θα τις εγκρίνω αλλά κάποιες νομίζω πρέπει να αναδιατυπωθούν είναι χρήσιμο να λάβουμε υπόψη μας την τροπολογία 165 της κυρίας Γκρέσλε για ένα συνολικό εξυγχρονισμό όπως προτείνεται από την ίδια. Αυτό είναι πολύ ένα πολύ καλό κείμενο και το συμπεριλαμβάνω στην έκθεση. Μία τώρα δυνητική τροπολογία συμβασμού και αυτό διότι πολλοί έχουν καταθέσει τροπολογίες για τη διαφάνεια. Και έχουμε προτείνει και μία τροπολογία οι πράσινοι έχουν καταθέσει μια τροπολογία και το ΕΛΚ και οι συντηρητικοί και οι μεταρρυθμιστές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε κάτι για το θέμα της διαφάνειας. Όχι να απορρίψουμε αυτά τα οποία έχει πράξει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρθηκαν στην αίτησή μας να υπάρξει απόλυτη αποκάλυψη όλων των δικαιούχων, αλλά δεν μπορούμε εδώ να παραγνωρίσουμε αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουμε στο θέμα αυτό της διαφάνειας. Θα ήθελα απλώ να προσθέσω στην ε, έγγραφη αυτή συμβιβαστική τροπολογία αυτή είναι και μια τροπολογία της κυρίας Μακοβέ ότι πρέπει να είναι αυτή η δήλωση σε μία από τις ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν παραγωγικά στη Λιθουανία υπάρχει μια βάση δεδομένων με διάφανα στοιχεία για το ποιος είναι αποδέκτης θα είναι πολύ δύσκολο για τον κύριο Στάς και τον κύριο Οντί να αντιμετωπίσει και να καταλάβει τι λέγονται, επομένως θα πρέπει να σε, σε μία από τις γλώσσες εργασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση αντικτύπου. Έχουμε πολύ καλές προτάσεις για τα θέματα αυτά. Και εγώ κατέθεσα μια τροπολογία για την ε, αξιολόγηση αυτή, ζητώντας να γίνεται με ανεξάρτητο τρόπο από ανεξάρτητους φορείς. Αυτή είναι η τροπολογία 12 και 13. Πρέπει να προσκαλέσουμε τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν τα κονδύλια τα οποία χρησιμοποιεί η Κομισιόν για εκθέσεις αντικτύπου σε ανεξάρτητους φορείς όπως παραδείγματος χάρη πιστεύματα και ιδρύματα. Γιατί ξέρετε ότι υπήρξαν πολλές φορές αμφιβολίες για τις εκθέσεις αντικτύπου που γίνονται από την Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούμε την ιδέα ενός ανεξαρτήτου φορέα ο οποίος θα προχωρήσει αυτές τις αξιολογήσεις. Η τροπολογία 109 του κ. Μπέλντερ που αφορά στο να αφήσουμε αυτό το θέμα στην κρίση της Κομισιόν δεν νομίζω ότι είναι συμβατή με μια τέτοια αντιμετώπιση και επομένως δεν μπορώ να τη δεχτώ. Εν τέλει, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ε, έγκρισης ή της αναβολής της απαλλαγής. Αυτό είναι το ουσιαστικό θέμα. Έχω δει τις τροπολογίες σας, τροπολογίες σας και ξέρετε ότι ο εισηγητής έχει καταθέσει και τις δύο τροπολογίες και για έγκριση και για αναβολή γιατί αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την απάντηση των αιτήσεων που έχουμε κάνει προς την Κομισιόν που έχουν καλυφθεί μόνο εν μέρη. Προς το παρόν και μετά από τη δεύτερη επιστολή πληροφόρησης από την Κομισιόν θα έλεγα ότι κατά βάση εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτό είναι το ενστικτό μου. Πρέπει να δώσουμε την ε, απαλλαγή. Υπάρχουν όμως δύο σημεία που είναι ακόμα εκρεμή. Βλέπω όμως ότι η Κομισιόν για ένα από τα δύο σημεία έχει αναφερθεί, έχει αναφέρει σαφώς ότι είναι ο έλεγχος απόδοσης, ότι οι πληροφορίες για το πώς το άρθρο 318 της Συνδίκης Λισαβόνας θα εφαρμοστεί, ότι είναι πληροφορίες που θα δοθούν στο Κοινοβούλιο, αυτό είναι κρυστάλλινα σαφές και κάτι άλλο το οποίο περιμένουμε από την Κομισιόν που είναι το βαθμολόγιο των κρατών μελών και διαφόρων ταμείων και αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πίνακα ο οποίος προς το παρόν είναι κενός ο πίνακας φαίνεται στο έγγραφο της Κομισιόν αλλά και ο οποίος πίνακας θα γεμίσει τουλάχιστον για το 2010 με αριθμητικά στοιχεία και από ό,τι, από ό,τι γνωρίζω η Κομισιόν για αυτή τη διαδικασία απαλλαγής θα λάβει υπόψη το βαθμολόγιο. Το βαθμολόγιο λοιπόν θα εφαρμοστεί ω ο αμέσως. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό εξασφαλίζει μια θετική διαφάνεια σε σχέση με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε λοιπόν πού τα πράγματα είναι καλά και πού δεν είναι καλά και επομένω εγώ πιστεύω πρέπει να περιμένουμε λιγάκι για αυτήν την ε, πληροφορία. Το ενστικτό μου μου λέει ότι έχουμε πετύχει ήδη αρκετά και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε την απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Εμείς πιστεύουμε ότι ούτως ή άλλως πρέπει να δώσουμε την απαλλαγή αλλά φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Αναφέρθηκε το θέμα του κανονισμού των υπαλλήλων, κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με τα θέματα τα οικονομικά που προκύπτουν από τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και τα δημοσιονομικά αυτά θέματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν πρέπει να έχουμε μια τέτοια τόσο επιφυλακτική στάση. Ξέρω ότι γίνεται και προσπάθεια lobbying πίσω από την πλάτη μου. Έχω κάνει πάρα πολλούς εχθρούς μέσα στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καθόλου μια συγκεντρωτική και παγιωμένη εικόνα για το πόσα άτομα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 50.000 περίπου αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πραγματικά απίστευτο και γι' αυτό τονίζω ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τα θέματα αυτά και άλλες τροπολογίες έχουν δημιουργήσει προβλήματα είναι χάρη το θέμα του flexi-time, του εύκαμπτου χρόνου εργασίας. Ε, υπάρχει εδώ μια διαφορετική αντιμετώπιση από μένα από ό,τι, όλα από ό,τι λέω κα, κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Υπάρχει και κάποιο λόμπι, λόμπινγκ εναντίον αυτής της ε, τροπολογίας, αλλά εγώ την υποστηρίζω γιατί θεωρώ ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να επανεξετάσουμε και να επεξεργαστούμε και να εξυγχρονίσουμε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και θα πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε χωρίς να ξέρουμε πόσο κοστίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια βάση αξιολόγησης. Και στην τελευταία διαδικασία απαλλαγή είχαμε αναφερθεί για το μηχανισμό της ε, τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, τη λεγόμενη μέθοδο για, την, ε, για τα θέματα αυτά και εκεί είχαν θεωρηθεί ότι δεν ήταν παραδεκτές οι τροπολογίες μας. Αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πιστεύω ότι και εδώ ως Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να τα δούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Βέλνερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα τόσο γλυκά σχόλια πολύ συμπαθητικό να μου πείτε δεν μου αρέσει τροπολογία σας, αλλά ευχαριστώ που την καταθέσατε. Πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ και εγώ που με ευχαριστείτε και χωρίς να σας αρέσει η τροπολογία μου. Ας περάσουμε όμως στην ουσία. Είπατε κάποιο σχόλιο για την ε, τροπολογία 272 με την ε, πρόταση για διαγραφή. Εγώ πιστεύω ότι και χωρίς να διαφωνώ ουσιαστικά με τη νέα λογική για τις δαπάνες, τη θέσπιση ενός προϋπολογισμού ουσιαστικού κτλ. Διαφανώς. Πιστεύω ότι για να έχει όμως την αξία το κείμενο αυτό θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο γιατί δεν μπορώ να δεχθώ. Δηλαδή φανταζόμουν ότι ο καθένας θα διαφωνούσε Θα έλεγα δηλαδή τι, πρακτική εφαρμογή έχει αυτό που λέγεται για εξασφάλιση πλήρους υποχρεώσεως λογοδοσίας στις δαπάνε κτλ. τα Στην αυτό δεν επιδιώκουμε. Όλη αυτή η διαδικασία αυτό δεν έχει σε στόχο. Χωρίς να λέω ότι είναι λάθος δηλαδή. Θα ήθελα κάποιο συγκεκριμένο. Και τώρα για κάτι που θέλω να συστήσουμε. Έχω κάνει το, το σφάλμα να φέρω τις τροπολογίες μου με, τα, με τη δική μου αρρύθμιση. Ασφαλώς θα ξέρει όμως ο γιατί σε τι αναφέρομαι. Ε, και εσύ είναι λάθος το νούμερο. Το θέμα των υπογραφών. Ποιος υπογράφει τις δηλώσεις, τις εθνικές δηλώσεις και γενικά ποιος υπογράφει. να επανέλθουμε στο θέμα αυτό που λέει θα υπογράφεται από τον Υπουργό shall be signed. Θα έλεγα κατά προτίμηση να πω, χωρίς αυτό να θέλω να μετατραπεί σε μια ε, γιατί δεν θέλω ε, να αποτελέσει αυτό μια δικαιολογία για εκείνους που δεν θέλουν να δεχθούν την υποχρέωση για υπογραφή και να πούνε αν δεν μπορεί πάντα να υπογραφεί Υπουργός, καλύτερα να μην υπογραφεί ποτέ. Όχι, θα ήθελα ε, να υπάρχει αυτή η προτίμηση και σε όλα τα κράτη-μέλη, έστω και αν δεν μπορούν πάντα να, υπογράφουν οι ίδιοι υπουργοί, να υπάρχει υποχρέωση για υπογραφή. Γι' αυτό θα έλεγα να μην δώσουμε ε, επιχειρήματα σε όσους θέλουν να αποτρέψουν ε, μια τέτοια επέμβαση. Αυτό. Αλλά λίγο πολύ αυτό το προτείνω σε όλο το κείμενο. Για την κυρία Γκρέσλε και τον κύριο Χατζημαρκάκη που και οι δύο αναφέρθηκαν στο κανονισμό του προσωπικού. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας στην έκθεση και με τόσο έχετε γράψει μέσα. Εκεί που πραγματικά διαφωνώ είναι το κείμενο που προτείνεται για το προσωπικό. Η προοπτική δηλαδή, που τουλάχιστον εγώ ερμηνεύω από το κείμενο, σαν να λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα για ορισμένα κράτη-μέλη, σε ορισμένα κράτη-μέλη η σταδιοδρομία του ε, υπαλλήλου δεν είναι αρκετά ελκυστική κτλ. Εγώ τουλάχιστον από τη σουηδική μου προοπτική θα έλεγα ότι ο κόσμος στη Σουηδία θεωρεί πως είναι μάλλον καλό πακέτο. η σταδιοδρομία αυτή. Και εάν είναι καλή προοπτική η σταδιοδρομία του ευρωιπαλληλου για ένα Σουηδό, σε ποια χώρα δεν είναι καλή και χωρίς να είμαι ειδικό, γιατί πολιτικό είμαι στη τελευταία ανάλυση, αλλά από όσου γνωρίζω εγώ προσωπικώ ε, στα θεσμικά όργανα και αντίστοιχα τους υπαλλήλου στην ε, Εθνική Δημόσια Διοίκηση, δεν μπορώ να πω ότι οι υπάλληλοι εδώ ε, περνάνε και άσχημα. Δεν μπορώ δηλαδή να δεχθώ ότι είναι δύσκολο να προσλάβουμε τους αρίστους. Δεν συμφωνώ με αυτό και γι' αυτό τροποποιώ και την διατύπωση. Επίσης, βλέπω κάποιο κείμενο για ένα φύλλο πορείας που ζητάτε για τις ε, δηλώσεις, εθνικές δηλώσεις και ε, το πώς θα ε, γίνει αυτή η δουλειά, πώς δηλαδή θα δώσουμε τη λύση. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να έχουμε μια διατύπωση που να μιλάει για τις εθνικές δηλώσεις και το ότι θα πρέπει να περιέχουν. Αλλά εκεί που διαφωνώ είναι η προθεσμία στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει μια εθνική δήλωση από κάθε κράτος μέλος συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ε, δύσκολο μου φαίνεται να ζητάμε μέσα σε μια χρονική στιγμή συγκεκριμένη όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ε, πράξει το ίδιο πράγμα όταν η Επιτροπή δεν μπορεί να τα ενημερώσει. Και θα ήθελα να δω και πώς μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Και ένα άλλο σημείο που βρίσκω θετικό, είναι και το καλύτερο της έκθεσης για την απαλλαγή. Είναι το σχετικό με την άρση των πληρωμών και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το ε, μέσον αυτό, το εργαλείο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο όταν κάποιο ε, εισπράττει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τα χρησιμοποιεί σωστά να έχει και τη σχετική κύρωση. Αλλά ίσω να μην ήμουν και. ίσω να παραήμουν ε, αισιόδοξο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να περιμένει δηλαδή να ε, βγαίνει σαν αλγόριθμος από ένα κομπιούτερ ε, αυτό το σύστημα. Αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προσμετρήσουμε το ε, πώς ε, εφαρμόζονται οι κανόνες. Άρα, αυτοματοποιημένα μεν, αλλά με κάποιο τύπου ε, επί, εποπτεία θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα. Και κάτι άλλο. Πρέπει να πω ότι εξεπλάγει μένα, αλλά δεν το περίμενα από την έκθεση, τον άρχισα να τη διαβάζω. Το βλέπω σε επιτομέρειες με τι τροπολογίες μόνο. Ότι δηλαδή ε, φαίνεται πως τα περιφερειακά ταμεία οι λογιστές υπογράφουν, λένε όλα καλά Α, ναι, υπηρεσίες πληρωμής. Και μετά σημειώνουμε ότι μάλλον δεν έχουν κάνει υπόψη τους, τους κανόνες βάσει των οποίων υπογράφουν. Υπογράφουν δηλαδή, ε, υπογράφουν έγκριση κάποιων ποσών τα οποία κακώς έχουν καταβληθεί. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να γίνεται η κατάρτιση. Πιο σωστά. Πολύ ωραία. Αλλά να σα πω, η μητέρα μου ίδια είναι λογιστρία. Δουλειά τη δεν είναι να ξέρει του κανόνε. Και εκείνη και κάθε λογιστή δεν έχει την ευθύνη. Κάθε λογιστή να ξέρει ποιου κανόνε εφαρμόζει. Και όταν βάζει την υπογραφή του και λέει ότι όλα έχουν γίνει ε, νομότυπα, ε, πρέπει να ξέρει ποιο είναι ο νόμο πάνω στον οποίο στηρίζεται αυτή η έγκριση, η επιβεβαίωση. Εγώ θα έλεγα, χωρί να ξέρω ακριβώ ε, τι θα πρέπει να, πώ ακριβώ θα πρέπει να το πούμε, ότι πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να λέμε ότι θα τους ε, εκπαιδεύουμε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Εάν μπορούμε να το διευθυντήσουμε κάποιον όλο τρόπο, πολύ ευχαριστώ να αποσύρω την ε, τροπολογία. Αλλά εν θεωρώ ότι είναι δουλειά τους να ξέρουν τους κανόνες. Τουλάχιστον έτσι το πρόξοφλο εγώ. Και για τους τριμερείς διαλόγους μεταξύ Προέδρου Επιτροπής, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Πολύ καλό. Αλλά ε, δεν νομίζω ότι η συνθήκη ε, επισημαίνει ε, ε, συγκεκριμένα τα πρόσωπα ή τους, ε, τη, τη, θέση αυτή ότι αναφέρεται σε προέδρους δηλαδή και ότι μάλιστα αν δεν το πράξουν αυτό οι πρόεδροι θα έχουν και σαν συνέπεια ε, μήνυσεις κτλ. Για όργανα μιλάει η συνθήκη. Και, εν το, το βασικό είναι να κάνει ο καθένα τη δουλειά του. Ε, το να λέμε ότι πρέπει να είναι παρόν το συγκεκριμένο πρόσωπο που εκπροσωπεί το θεσμικό όργανο και ότι η απουσία θα έχει σαν συνέπεια, απουσία σε συνέπεια την άσκηση μήνυση τη βάρο του, δεν νομίζω ότι συνάδει κανένα τη συνθήκη. Ευχαριστώ πολύ, Ιβάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω πολλά να πω γιατί νομίζω ότι είχαμε μια θαυμάσια σχέση με τον κύριο εισηγητή, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την εκθεσή του και για την πολύ καλή επικοινωνία που είχε με τους κοιόδης εισηγητές για όλες τις διάφορες πτυχές της έκθεσής του που πρέπει να τύχουν περαιτέρω διευκρίνησης. Η σχέση με την Κομισιόν ήταν επίσης πολύ καλή και σε όλε τι διαπραγματεύσει εμεί προσπαθούμε να επιτύχουμε ό,τι είναι δυνατόν να επιτύχουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε τα πάντα, αλλά η Κομισιόν έχει κρατήσει μια επικοδομητική στάση και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα με αυτή την έκθεση για μια καλύτερη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Ταμείων στο μέλλον. Υπάρχει ένα σημείο <clears throat> δυσαρέσκειας ακόμα για μένα. Οι εθνικές δηλώσεις διαχείρισης θα πρέπει να υπογράφονται από ένα υπουργό, από κάποιον που να έχει πράγματι και κάποια υπευθυνότητα στα θέματα αυτά. Γιατί αλλιώς οι αξίες αυτών των δηλώσεων δεν είναι ιδιαίτερες. Η αξία αυτών των δηλώσεων εξαρτώνται από το επίπεδο στο οποίο υπογράφονται. Αν είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει μεγάλη σημασία, τότε αυτή η δήλωση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει ικανοποιητικό χαρακτήρα. Και οι πληροφορίε αυτέ δεν θα είναι εμπεριστατωμένε αν δεν γίνεται σε υψηλό επίπεδο υπογραφή. Γι' αυτό έχει σημασία λοιπόν το ποιο αναλαμβάνει τα θέματα αυτά. Θέλω να σταματήσω εδώ, όπω είπε και ο κ. Χατζημαρκάκη. Εμεί έχουμε συμφωνήσει στο, στη διαδικασία για τι τροπολογίε παρά το γεγονό ότι είναι πολλέ. Η κυρία Αγιάλα και Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να λάβει υπόψη του ο κύριος Χατζημαρκάκης τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει για την τελική, τελικό κατάλογο ψηφοφορίας. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα άγρια λόμπι που είναι ελοχεύοντα πίσω από την πλάτη της κυρίας Γκρέσλε, αλλά βέβαια αν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο κάποια καταπάτηση χωραφιών άλλων επιτροπών, αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά θα δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ έχω σταθεί συνδικαλίστρια στο παρελθόν για τα θέματα του προσωπικού και μπορώ να κατανοήσω ορισμένα από αυτά τα οποία ελέγχθηκαν και συμφωνώ για ορισμένα τα οποία ελέγχθηκαν και θα δούμε τι θα προτείνει ο εισηγητής της προτάσεις ε, ε τροπολογίας αλλά για ορισμένες από τις προτάσεις της κυρίας Γκρέσλε για να τροποποιήσουμε κατα, καταρχήν το εβδομαδιαίο βάρος εργασία των υπαλλήλων, αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ένα επωφελή χαρακτήρα, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τη δική σας χώρα και τη δική μου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν είμαστε προοδευτικοί ή όχι για τα θέματα αυτά. Και επίσης θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Γκρέσλερ σε ό,τι αφορά το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση των εθνικών υπαλλήλων. Και θα έπρεπε να σκεφτούμε ποιος είναι ο υπάλληλος, ο μέσος υπάλληλο. Αν δείτε αυτούς οι οποίοι ζουν στις Βρυξέλλες δεν ζουν στον καλύτερο των δυνατών κόσμων. Και μια τροπολογία η οποία επίσης νομίζω ότι πρέπει να την ξανασκεφτεί η κυρία Γκρέσλε είναι η 163 υπάρχουν κάποιες φήμες που περιστρέφονται γύρω από αυτήν και δεν μου αρέσει να δουλεύουμε επί τη βάση φήμων αλλά το να ζητήσουμε όπως λέει η τροπολογία ότι υπάρχουν νέοι οι νέοι πάλι είναι νέοι καταρχήν ότι υπάρχουν νέοι πάλι ότι μπήκαν μετά από τη διεύνηση και οι οποίοι ανήκουν ή ανήκανε σε υπηρεσίες, σε μυστικές υπηρεσίες των ε, πρώην κομμουνιστικών κρατών και ότι πρέπει να δώσουν μια δήλωση πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα, αυτό μου φαίνεται ότι είναι κάτι το ολοκληρωτικό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση που ήταν η Γερμανία το 1989 και δεν μπορούμε εμείς να ακολουθήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι και από τους κοινοβουλευτικούς μας μπορεί να αναφερθεί ότι ίσως και αυτοί θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή να κάνουν μια αντίστοιχη δήλωση πριν κατέβουν στις εκλογές. Επομένως, είναι ένα θέμα το τι κοστίζει η Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία, αυτό μπορούμε να το θέσουμε, αλλά τροπολογίες οι οποίες έχουν το περιεχόμενο αυτό που ανέφερα, νομίζω ότι δεν είναι πραγματικά παραδεκτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γκρέτ. Ines, du redest immer so schnell. Da kommt immer der Dolmetscher nicht Ich wollte nur sagen, die ναι, τα είπατε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η τροπολογία 73, εκεί που μιλάμε για ένα μηχανισμό επαλήθευσης screening για τους ε, μελλοντικούς υπαλλήλους, με μια διαδικασία επαλήθευσης και δηλώσεων ότι δεν ήταν μέλη μυστικών υπηρεσιών. Και αυτό το λέω γιατί μου το έχουν ζητήσει και οι προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων από τη Γερμανία. Το Δεκέμβριο του 2010 έγινε μια μελέτη στη Βουλγαρία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ζήτησε από τους δικούς του να του πούνε πόσοι από αυτού είχαν διατελέσει μέλη μυστική υπηρεσία και περίπου 300 απάντησαν θετικά. Άρα πρέπει να υπάρχει κάποιο μηχανισμό. Δεν θα το πίστευα εγώ ίδια ότι θα είχαμε τέτοιου είδους κλίμακες. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι γεγονός αυτό. Διαπιστώθηκε και χωρίς να θέλω να αμαυρώσω κανενός τη φήμη, υπάρχει αυτή η μελέτη και πιστεύω ότι και τα κράτη-μέλη τα ίδια θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Άρα κάποια, κάποιου τύπου ε, δήλωση, επαλήθευση θα πρέπει να υπάρχει και χωρί να περιμένουμε πολύ, γιατί διαφορετικά θα καταρρεύσει η Ευρώπη και λύση δεν θα έχουμε βρει ακόμα. Αν δεν υπάρχουν άλλε ε, ερωτήσεις, τοποθετήσει. ο κύριος Κάλφιν όμω. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, μια και το ανέφερε η κυρία Γκρέσλι, υπήρξε μια περίπτωση στη Βουλγαρία. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σας απαντήσω. Υπήρξε λοιπόν. Ξέρετε ότι έχουμε και μια νομοθεσία στην Βουλγαρία η οποία έχει να κάνει με την ε, προσφορά υπηρεσιών στην ε, ε, μυστική υπηρεσία του προηγούμενου, του παλαιότερου καθεστώτος, του κομμουνιστικού καθεστώτος. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τη δραστηριότητα και την, την έρευνα που έκανε το Υπουργείο των Εξωτερικών. Πολύ σωστά είπατε ότι ήταν περίπου 200 αυτοί που απάντησαν, αλλά ήταν η περίοδος των, της τελευταίας 20 ετίας, δηλαδή μετά το 90. Αυτό δεν αφορά τους 600 διπλωμάτες που τώρα υπηρετούν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είναι από αυτούς 600-200 πρώην ε, μέλη της μυστικής υπηρεσίας. Η μελέτη δείχνει ότι τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχαν 200 στο διπλωματικό σώμα συνολικά που υπηρέτησαν και πιο πριν βέβαια άλλοι. Άρα είναι πολύ διαφορετικές οι αναλογίες από αυτό που παρουσιάζεται, κυρία Γκρέσλε. Κύριο Χατζημαρκάκη. Ναι, και αρχίσαμε τη συζήτηση αυτή. Την τροπολογία 173. Θα βρούμε μια λύση, φαντάζομαι. Θα το ρυθμίσουμε. Όμω πιο κρίσιμη, και αρχίζω με τα όσα είπε η κυρία Γκρέσλε, είναι η τροπολογία. Είναι το σημείο που ξεκινάμε με την 170 εκεί που γίνεται λόγος για το άρθρο 56 του κανονισμού προσωπικού και γίνεται μια προσπάθεια να συζητήσουμε το πώς διαμορφώνεται η λειτουργία των υπαλλήλων. Βεβαίω και μπορούμε να το πράξουμε. Η Επιτροπή μας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό και δεν είμαι 100% κατά τις δικές σας τροπολογίες. Θα το αφήσω στην κατασυνέδηση ψήφου. Αλλά η επόμενη τροπολογία, εκεί όπου καλείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, απαλείψει πεπαλαιωμένες ε, διατάξεις περί επιστροφής των εξόδων κτλ. Ε, θα ήθελα να ε, τη δούμε με τρόπο διαφοροποιημένο και μάλιστα σε τμήματα και σε δεύτερο τμήμα. Εκεί που λέτε να προσαρμοστούν οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αντίστοιχες αλλαγές στο προσωπικό των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, δεν είναι η θέση του εκεί. Στην επόμενη τροπολογία. για την ε, είσοδο στην ε, σταδιοδρομία στο επίπεδο AD5. Μπορώ να το δεχθώ και όπως επίσης και το θέμα της παροχής υπηρεσιών σε ε, συγκεντρωτικά καθεστώτα. Δέχομαι λοιπόν ως ιδέα τις τροπολογίες όπως βλέπετε στο σύνολό τους. Για τις 50 τροπολογίες του κύριου Φιέλναρ, για τις οποίες ήμουν ευγνώμων όπως είπα, θα ήθελα να τους δείξουμε μια ματιά. Εκεί που λέτε λοιπόν ότι πρέπει να διαγραφεί η απέτηση για την ασαφή διατύπωση. Θα σας καλούσα να ρίξετε μια ματιά στην επιστολή του κύριου Σέμετα. Η οποία μπορεί να σας ξαφνιάσει, γιατί ίσως δεν είναι εκ πρώτης όψεως, αλλά στην ουσία είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν περίμενα τόση σαφήνεια εγώ από την απάντηση αυτή και γι' αυτό δεν πρέπει να απαλληφθεί το σχετικό κομμάτι. Είναι πολύ καλή λοιπόν η απάντηση. Για την πρότασή σας οι υπουργοί των εθνικών κυβερνήσεων να υπογράφουν κατά προτίμηση την δήλωση. Πολύ ευχαριστώ να συμφωνήσω για το προσωπικό έδωσα τι απαντήσει μου. Την πρώτη ερώτηση. Για το φύλλο Η τροπολογία σας στόχο έχει να νερώσει τρόπον την το κείμενο. Ο κύριο Μπέλτερ ζητάει ότι μέσα απαιτεί σε μια δική τροπολογία ότι ε, σε δύο χρόνια αμέσω πρέπει να έχουμε τον υπουργό κτλ. Ε, γι' αυτό ακριβώ το λόγο, όπω είπα και στην αρχή, πρέπει να εμείνω στην δική μου θέση που υποστηρίζει και ο κύριο Σίβαν και τον ευχαριστώ. Για τον αυτοματισμό, τη, ρο, τη ρομποτιά που λέτε, έχετε δίκιο. Εγώ πήρα κάποιες από τις τροπολογίες σας και κάποιες από των σοσιαλιστών Οπότε το κείμενο με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί και σας ευχαριστώ. Για την ε, κατάρτιση των λογιστών των διατακτών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Κομισιόν ήδη στην πρώτη της επιστολή έχει δώσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα πρέπει να γίνεται η εκπαίδευσή τους γιατί γίνονται συνέχεια αλλαγές στο σύστημα. Και οι Σουηδοί λογιστές θα πρέπει και αυτοί να το ξέρουν Υπάρχουν όμως μερικά κράτη-μέλη, ιδίως στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης, όπου τα μέτρα εκπαίδευσης είναι κάπως ελλειπή ίσως. Μια χώρα που είναι 30 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται πολύ μα πολύ εκπαίδευση για τους λογιστές της. Γι' αυτό εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόταση που βρίσκεται στην πρώτη επιστολή της Κομισιόν για το πού πρέπει να εκτελ... πότε και πού πρέπει να υπάρχει κατάρτιση αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτό δεν έχει γίνει επαρκώς στο παρελθόν, τουλάχιστον στο επίπεδο που θα θέλαμε όλοι. Σας ευχαριστώ επίσης και για τις διευκρινήσεις σας για το ποιος θα πρέπει να πηγαίνει στο δικαστήριο. Θα το ξανακοιτάξουμε. Γιατί η συνθήκη μαζί με τους με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, γιατί από εκεί έρχεται το, ο κανονισμός. Λέει ότι σε καταστάσεις όπου υπάρχουν θεσμικά προβλήματα, και το συζητήσαμε αυτό χθες, όταν μιλούσαμε για την απαλλαγή του Συμβουλίου, είναι οι τρεις πρόεδροι οι οποίοι πρέπει να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ τους. Αλλά ίσως πρέπει να το ξανακοιτάξουμε και να το αναφέρω στον κατάλληλο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω και τους κυρίους ε, από τη Σοσιαλιστική Ομάδα, την κυρία Γιάλα Σέντε και τον κύριο Κάλφιν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Και ελπίζω ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας που θα συζητήσουμε με τους κοιόδη συζητητές την 5η 9 ώρα το πρωί, όταν κάνουμε την τελευταία αυτή επεξεργασία, θα σας βρει όλους σύμφωνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Χατζή κάκι. Τέλειωσε η δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Συνεχίζουμε με τους συντονιστές και χαιρετούμε τους υπόλοιπους.